Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht immer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, μας πιέζει ο χρόνος γιατί έχουμε βαριά ημερήσια διάταξη και σήμερα και αύριο. Παρόλη τη μικρή σχετικά προσέλευση θα αρχίσουμε. Το σχέδιο ημερήσια διάταξης θα εγκριθεί αν, αν δεν διαφωνεί κανεί, όπως και δεν διαφωνεί. Τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και πάλι αν δεν διαφωνήσει κανείς. Είναι της 26ης Μαρτίου και πάλι δεν βλέπω διαφωνίες και αντιρρήσεις. Πάμε λοιπόν στο σημείο 3 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κίρκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τη γραμματεία της Επιτροπής Μεταφορών και τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Λάβαμε 139 τροπολογίες, συμφωνήσαμε σε 8 συμβιβασμούς, οι οποίοι έχουν τη στήριξη των πολιτικών ομάδων που συμμετείχαν. Τις ευχαριστώ. Θεωρώ ότι με τροπολογίε το κείμενο έχει εμπλουτιστεί και φωτίζει επαρκώ όλε τι παραμέτρου του πολιτιστικού τουρισμού, τι οποίε θα ζητήσουμε από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία, που είναι επί τη ουσία αρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα να συμπεριλάβει. Να τονίσω εδώ ότι όπω εξήγησα και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε του Κιώδη, ο λόγο που κάποιε τροπολογίε έχουν αρνητικό πρόσημο είναι είτε γιατί ήδη υπάρχουν μέσα στο κείμενο, είτε γιατί αναφερόντουσαν σε θέματα πολιτισμού και αυτά θα περιληφθούν στην έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού ή σε θέματα τουρισμού και θα καλυφθούν από την έκθεση της δικής μας Επιτροπής για τον τουρισμό και όχι στις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα διακυβεύματα που δημιουργούνται από τις συνεργασίες των δύο. Προσπαθήσαμε δηλαδή να κρατήσουμε ένα κείμενο με προτάσεις που αφορούν πολύ συγκεκριμένα τον πολιτιστικό τουρισμό, τον οποίο και αυτό θεωρώ πως το καταφέραμε με τις τροπολογίες των συναδέλφων. Η γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις, όπως τόνωση του πολιτιστικού τουρισμού σε αγροτικέ, ορεινέ, παράκτε και νησιωτικέ περιοχέ, που προσφέρουν άθικτο φυσικό περιβάλλον και τοπία, παραδοσιακό πολιτισμό, τοπικά προϊόντα, γαστρονομικέ παραδόσει και γνησιότητα. Η ενίσχυση σε αυτέ τι περιοχέ αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την τοπική ανάπτυξη. 2. Λήψη μέτρων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την εξασφάλιση ενό επαρκού ρυθμιστικού πλαισίου των επιχειρήσεων, ιδίω των μικρομεσαίων και των νεοειδρυθισών, που ενεργοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. 3. Αξιοποίηση των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό, διαφάνεια και πιο ανοιχτή προσέγγιση εκ μέρου τη Επιτροπή σχετικά με την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προώθηση τη πολιτιστική κληρονομιά. 4. Διασφάλιση αηφόρου και υπεύθυνου τουρισμού που θα ανταποκρίνεται στι ενδεχόμενε αρνητικέ επιπτώσει των διαρθρωτικών αλλαγών που προκαλεί ο τουρισμό και στου κινδύνου που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά λόγω μαζικού τουρισμού αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη ψηφιοποίηση τη πλούσια πολιτιστική κληρονομιά τη Ευρώπη ω μέσο για την προώθηση του μοναδικού πολιτιστικού τη πλούτου παγκοσμίω. Έκτο, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων όπω είναι οι ευρωπαϊκέ πολιτιστικέ διαδρομέ. Και εδώ να κάνω μία παρένθεση και να επισημάνω την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής για το Iron Curtain Trail και πώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στη διάνοιξη καινούριων διαδρομών στην Ελλάδα. Έβδομο, ανάπτυξη βιώσιμων διατροπικών υποδομών και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα για τη βελτίωση τη προσβασιμότητα εν γέννη και ιδίω των απομακρυσμένων τουριστικών προορισμών. Όγδο και τελευταίο, διευκόλυνση προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίε ή χαμηλή κινητικότητα, καθώ και σε οικογένειε με χαμηλά εισοδήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πολιτιστικό τουρισμό αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του ευρωπαϊκού τουρισμού χάρη στην πλούσια πολιτιστική, καλλιτεχνική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά, τους φυσικούς πόρους, τη γεωγραφική θέση, την ποικιλία των τοπίων της. Όμως η οικονομική κρίση έχει στερήσει κονδύλια από ένα τομέα που έχει πληγεί περισσότερο από τις περικοπές, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη, παραμέληση και υποβάθμιση πολύτιμων πολιστικών αξιοθέατων, σε βάρος της κοινωνίας και του τομέα του τουρισμού. Κλείνοντα, θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία των συνεργειών μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού και τη συνεισφορά του στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση είναι πολύ μεγάλη. Ελπίζω οι προτεραιότητέ μα να είναι σαφεί στην έκθεση και να ληφθούν υπόψη από την κατουσία αρμόδια επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι παρόντες όλοι οι σκιώδεις συζητητές. Ποιος θέλει το λόγο, ε, Πιέζει ο χρόνος βέβαια. Καριμαντελή. Ε, η... Πρώτα έχει το λόγο η κυρία Καυσίσκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση ψηλής ποιότητας και πολύ καλή έκθεση γενικότερα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συνένεση τελικά. Είχαμε 139 τροπολογίες. Ο εισηγητής όπως και οι σκιώδεις έφτασαν σε 8 συμβιβασμούς και μία προφορική τροπολογία και την υποστηρίζω γιατί έχει να κάνει με άτομα περιορισμένης ε, κινητικότητας και χαμηλόμισθους. Εργάστηκα για την έκθεση αυτή γιατί με ενδιαφέρει ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού. Το τονίσατε και εσείς αυτό. Εγώ προέρχομαι από το Ντουμπρόβνικ που έχει μεγάλη ε, πολιτιστική κληρονομιά και πλήττεται από μαζικό τουρισμό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διατηρήσουμε τον, την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά από την άλλη να μπορέσουμε να προσφέρουμε ε, ποιοτικό τουρισμό. Αυτό δεν αφορά μόνο την Κροατία, αλλά ολόκληρα την Ευρώπη. Συζητήσαμε επίσης πώς η Ευρώπη να γίνει ο πρωταρχικός προορισμός τουρισμού ανά τον κόσμο. Αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμο τουρισμό παντού στην Ευρώπη, θα πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά πρωτίστως. Πρόκειται για κληρονομιά των προγόνων μας και θα χρησιμοποιηθεί και από τα παιδιά μας, αφορά και τα παιδιά μας στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να πω και κάτι άλλο πολλές τροπολογίες που προήλθαν από το ΕΛΚ θα έπρεπε να θεωρηθούν ε, θετικές. Είπατε όμως ότι έχουν περιληφθεί στο κείμενο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να υποπτεύουμε τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού, να σκεφτούμε το, την αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλή ποιότητα. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική τομή στον τουρισμό. Εάν υπάρχει συνέργεια μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού, θα προωθήσουμε και την απασχόληση καθώς και τη διατήρηση του πολιτισμού μας. Δεν θέλουμε η ανάπτυξη του τουρισμού όμως να θέσει σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. Θα πρέπει να κάνουμε μία ιεράρχηση και να προβάλλουμε τις προτεραιότητές μας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή και αύριο θα φτάσουμε σε συνένεση πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Τόμας Πορέμπα. E, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω τις ευχαριστίες που εκφράστηκαν για τον εισηγητή διότι μας έδωσε μία πλήρη περιγραφή του θέματος και οι τροπολογίες που κατέθεσα και είδα ότι έχουν συμπεριληφθεί στις συμβιβαστικές εξ ονόματος των συντηρητικών κατατέθηκαν για να βελτιώσουν το κείμενο και χαίρομαι ιδιαίτερα που η εισηγητής τις δέχτηκε και τις συμπεριέλαβε για να μιλήσουμε όλοι μαζί για την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Ιδιαίτερα το σημαντικό για μένα είναι τα κεφάλαια, τα τμήματα που αφορούν τις ρίζες, τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης, που νομίζω ότι είναι η βάση των αξιών μας. Και άλλες τροπολογίες έχουν συμπεριληφθεί, ως πούμε, ό,τι αφορά την προώθηση του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού στο Μαυροβούνιο ας πούμε. Εγώ είμαι από ένα τμήμα της Πολωνίας όπου έχουμε περιοχές με πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και φυσικά θέλουμε να προωθηθεί ο τουρισμός και τοπικά γιατί υπάρχουν πολλά μνημεία που πρέπει να τα γνωρίσουν περισσότεροι. Άρα μεγαλύτερη πρόσβαση σε όλες τις περιφέρειες. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ορισμένα προγράμματα που τονίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό, τον πολιτιστική κληρονομιά και υπάρχουν και πολύ επικοδομητικά και βιώσιμα παραδείγματα από τα οποία να εμπνευστούμε και που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Εξ ονόματος των Δυτικών λοιπόν συγχαίρω ακόμη μια φορά τον εισηγητή για την εξαιρετική του γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρτίνα Δλαμπάγιο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, εξ ονόματος των φιλελευθέρων, να συγχαρώ τον εισηγητή και του σκιώδης. Ήταν πολύ αγαστή η συνεργασία, πολύ καλή δουλειά έχει κάνει και ο εισηγητής με τους συμβιβασμού και ε, πραγματικά ε, θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες για τις συμβουλές τους σε τέτοια θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποιον άλλο να ρωτήσουμε καλύτερο. Ε, χρειάζεται διασφάλιση, προστασία και προώθηση και διαφήμιση πολιτιστική μας κληρονομιά. Ε, πολλά τα είπαν ήδη οι συνάδελφοι, θέλω να ε, προσθέσω τα εξής τρία. Πρώτον, θα πρέπει να μειωθεί ε, το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μην υπάρξουν ε, αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία τους, στον τουρισμό και ε, στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό το έχετε βάλει στη συμβαστική τροπολογία 7 και ευχαριστώ. Επίσης, δεύτερον, η άμεση πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά στα κονδύλια. Ε, με περισσότερη διαφάνεια να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια αυτά ε, με διαφανή διαχείριση και διαφανή τρόπο και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει λόγο. Αυτά τα λέει ο Συμβασμός Υπαριθμών 8. Τρίτον, η διασυνοριακή ε, διασύνδεση θα πρέπει να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα ε, παροχής ε, εισιτηρίων, ενιαίο εισιτήριο και ενιαίο τρόπο προγραμματισμού των διακοπών των πολιτών για να διευκολύνεται αυτή η επαφή. Έχω όμως μία ανησυχία που αφορά τη μοναδική προφορική τροπολογία που έχει υποβάλει ο εισηγητής. Συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα. Για μένα όμως η διατύπωση οδηγεί σε σύγχυση. Πώς το συνδέεται με τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η προφορική τροπολογία, να γίνει πιο ε, σαφής και κατανοητή για όλους. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία που είχαμε και ε, για τα σχόλια μου που πήρατε υπόψη και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καρίμα Αντέλη. Ευχαριστώ εξ ε, της G. 11 θα ήθελα να πω ότι ευχαριστεί για την εργασία του εισηγητή και έχει επιτελεστεί πρόοδος ιδιαίτερα σε σχέση με τους συμβιβασμούς. Φύγεται ζητήματα τα οποία είναι ύψης της σημασίας ως προς την προσβασιμότητα υψηλής ποιότητας. Επίσης να λάβουμε υπόψη τις ορεινές περιοχές, τις παράκτιες ε, περιοχές, τα νησιά, ε, όλες τις γλώσσες και διαλέκτους και να τονίσουμε τις νέες τεχνολογίες, την πληροφόρηση και την επικοινωνία, όπως και τον προγραμματισμό ολοκληρωμένων ε, ταξιδιών Μας ενδιαφέρει να λάβουμε υπόψη τα περιφερειακά σχέδια και τα διασυνοριακά και μιλήσατε και για βιώσιμο τουρισμό στην εισήγησή σας. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλός για τον πλανήτη και για τις μελλοντικές γενές. Άρα στους συμβιβασμούς που προβάλλουμε. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το νέο τρόπο ανάπτυξης, ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας μέσα όπως ποδηλατοδρόμους, σιδηροδρομικά δίκτυα μέσα στα πλαίσια του τουρισμού και ιδιαίτερα ως προς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που έχουν κλείσει. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ό,τι προϋπάρχει και ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Για μας έχει μεγάλη σημασία η διαφάνεια στη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων και καλύτερη χρήση τους. Είμαστε ε, ικανοποιημένοι από πλευράς οικολόγων ως προς τους συμβασμούς και πιστεύω ότι θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ισαπέλα Δημότ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή όχι μόνο για την έκθεση αλλά και για τις τροπολογίες που δέχτηκε. Πρόκειται για θέματα που είναι πολύ σημαντικά και για τον τουρισμό. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε το, την πολιτιστική μας κληρονομιά γιατί περιορίζεται και ο τουρισμός. Θα πρέπει όμως να σταθούμε και στο θέμα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή σημασία η συνολική προσέγγιση της κληρονομιάς. Μας ενδιαφέρει η ταυτότητα, διότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία. Οι γλώσσες των μειονοτήτων, η πολυπολιτισμικότητα και ούτω καθεξής επίσης. Λάβαμε υπόψη τις ορεινές περιοχές, τις απομακρυσμένες περιοχές τις ε, περιοχές με νησιωτικό χαρακτήρα και ούτω καθεξής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι σε αυτές τις περιφέρειες ε, ε, δυστυχώς αποδυναμώνεται ο πληθυσμός, μεταφέρεται αλλού και άρα ερημώνουν αυτές οι περιοχές μιλήσαμε και για πρακτικά ζητήματα, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών και έχει σημασία οι πληροφορίες να υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες για να έχουν πρόσβαση όλες τις πληροφορίες αυτές. Ευχαριστώ κυρία Μαρία Γκραπίν. Εντάχει, θα πρέπει να σας ε, ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον εισηγητή καθώς και όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Μία ανησυχία θα ήθελα να εκφράσω. Πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη υπό την οπτική γωνία της ανάπτυξης του τουρισμού. Έχει σημασία να δούμε την τροπολογία 12. Στην ουσία αντιτίθεται σε αυτό που προτείνουμε. Βεβαίως υπάρχει ο μαζικός τουρισμός, τον οποίο αν δεν διαχειριστούμε σωστά μπορεί να πλήξει την ε, κληρονομιά μας. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τον ε, τουρισμό. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να κινηθούμε προς τον τουρισμό των πλουσίων δεν πρέπει να ε, αναχαιτήσουμε τον μαζικό τουρισμό. Πιστεύω ότι η τροπολογία υπαριθμών 12 αποκλείει τον μαζικό τουρισμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην τουριστική βιομηχανία. Θα ήταν σκόπιμο να αρκεστούμε στην αρχική διατύπωση της τροπολογίας 12. Δηλαδή να μιλήσουμε για ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες, αλλά να μην, μιλάμε για, να μην έχουμε αυτή την αρνητική προσέγγιση. Ευχαριστώ κύριο Σκύρικος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τους ομιλητές σήμερα. Ήταν μια ένδειξη του πόσο ενδιαφέρον ήταν ο διάλογος που διατρέξαμε και πόσο είναι κοινά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε ε, στο θέμα του πολιτισμικού τουρισμού. Ε, όπως για παράδειγμα το Ντουμπρόβνικ που είναι ένα πετράδι, αλλά για να παραμείνει πετράδι πρέπει ο μαζικός τουρισμός ο οποίος κατευθύνεται προς τα εκεί να μπορέσει να διοχετευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέψει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης γιατί μετά δεν θα έχει περιεχόμενο ακριβώς ο στόχος. Και αυτό είναι κάτι που ε, το έθιξε και η κυρία Γκραπίνη είναι όντως ότι ε, προχωράμε προς μια κατεύθυνση που ο τουρισμός γίνεται όλο και πιο μαζικός και μιλώντας για αύξηση του αριθμού των τουριστών προσανατολιζόμαστε στο να φέρουμε όλο και περισσότερους ε, τουρίστες στα διάφορα μέρη. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε τον μεγάλο αριθμό. Όχι να σταματήσουμε την ροή που είναι και κάτι δύσκολο έτσι όπως γίνεται και η ανάγκη του, των, της ανάπτυξης οδηγεί προ την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το πλήθο των τουριστών. Εμεί έχουμε στην Ελλάδα το πράγμα τη Σαντορίνη, όπου δέχεται δεκάδε κρουαζιερόπλια κάθε μέρα και πραγματικά βουλιάζει το νησί. Η απάντηση δεν είναι να μην έρχονται τα κρουαζιερόπλια, να κάνουμε τέτοιου τρόπου κατανομή μέσα στον χρόνο που το έχουν, συζητήσει, έχουν ζητήσει και οι ίδιοι οι τουριστικοί πράκτορε, ώστε να μπορέσουν να έρθουν οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά ακριβώ να απολαύσουν αυτά που δίνει το νησί και την, ε, το φυσικό τοπίο, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά με ένα τέτοιο τρόπο που θα προσλάβουν αυτό για το οποίο έρχονται. Άρα είναι θέμα της διαχείρισης και όχι της άρνησης φυσικά. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους άλλους ομιλητές. Όντως η προσβασιμότητα είναι ένα μεγάλο, όπως είπε ο κύριος Πορέμπη, η προσβασιμότητα και των μνημείων, το οποίο είναι και, και άγνωστα σε πολλές πλευρές και πρέπει να προβληθούν, αλλά ακριβώς πρέπει να υπάρχει τρόπος να φτάσεις εκεί. Η σημασία των μικρομεσαίων που μας τόνισε η κυρία Δελάγιοβα. Ε, διατρέχει όλο το κείμενο ότι αυτό που πρέπει να στηριχθεί είναι ακριβώς οι τοπικές κοινωνίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του, της τουριστικής ανάπτυξης και αυτές πρέπει να τις διευκολύνουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και φυσικά ε, μέσα στο κείμενο το διαπερνάει και η ανάγκη να μην μιλάμε για λίγους προορισμούς, αλλά να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τους πιο ε, απομακρυσμένους, είτε είναι σε ορεινές περιοχές, είτε σε μακρινά νησιά, γιατί η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό το διαφορετικό, αυτές οι πάρα πολλές πλευρές, αυτό είναι το μεγάλο όπλο μας σαν ε, Ευρώπη πρώτος τουριστικός προορισμός και αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε. Και φυσικά όλοι οι τρόποι οι οποίοι διατηρούν ε, το φυσικό περιβάλλον, διατηρούν τα, τα, χωριά, αυτό που είπε ε, η κυρία Ντέλη από τους Πράσινους, οι ποδηλατόδρομοι, τα, τα μονοπάτια, όλοι οι τρόποι δηλαδή που μπορεί ο τουρίστας, ο επισκέπτης να νιώσει έναν ένας με τη φύση είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προωθηθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι και τους ομιλητές σήμερα αλλά και τους σάντους που κάναμε πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω αύριο να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί ψηφίζουμε την έκθεσή σας. Ωραία. Ε, πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Παρουσίαση της κοινή έκθεσης προόδου των Ευρωπαίων Συντονιστών. Καλωσορίζω τον Ματιό Εγκρό εδώ και τον Πατ Κόξ. Πάρα πολύ γνωστή και οι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Όπως γνωρίζετε, το έτος 2014 ήταν αφεταρία για τα ε, νέους ε, διαδρόμους με το Connecting Europe και το TNT, τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Ματιού Γκρός λοιπόν και Πατ Κόξ από κοινού θα μας παρουσιάσουν την κοινή έκθεση προόδου για τα προγράμματα αυτά, καθώς επίσης και το βασικό δίκτυο και τους, ε, τις λεγόμενες λεωφόρους της θάλασσας. Θα ξανάρθουν ε, για τα επιμέρους, μην τους ρωτήσετε γι' αυτά. Τώρα θα μας παρουσιάσουν την ενδιάμεση έκθεση και των 11 συντονιστών. Πριν τους δώσω το λόγο θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 ε, ε, του κανονισμού TNT και οι 11 συντονιστές θα προσκληθούν εδώ έτσι ώστε να μας παρουσιάσουν επιμέρους ο καθένας την ετήσια έκθεσή του. Και θα σας ξαναδούμε σας δύο και τότε. Αυτές οι εκθέσεις ε, θα παρουσιαστούν εδώ στην Επιτροπή μας από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος και θα πρέπει να φροντίσω εγώ να τηρήσουμε το χρόνο μας. Σήμερα όμως θα μας απασχολήσει η ενδιάμεση κοινή έκθεση για το 2014 και των 11 συντονιστών. Πριν από 15 μέρες τη λάβατε όλοι ηλεκτρονικώς, την έχουμε και σήμερα εδώ και θα δώσω το λόγο και στους δύο, δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει, ο Πατ Κόξ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Mr. Uh, Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Είναι μεγάλη η δονή που αισθάνομαι καθώς και του κυρίου Γκρός να βρισκόμαστε μπροστά σας σήμερα. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαμε ως συντονιστές να σας μιλήσουμε από τις ευρωεκλογέ και μετά. Και είναι η πρώτη φορά που σας μιλώ εγώ, εσάς κύριε Πρόεδρε, ως Προέδρο. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε μια κοινή αποτίμηση εξ και των 11 συντονιστών. Όχι με τις συγκεκριμένες αναλύσεις που είπε ο Πρόεδρος. Αυτές θα γίνουν αργότερα σήμερα. Θέλουμε να σας πούμε τι έγινε κατά το πρώτο έτος των διαδρόμων αυτών από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013 ενέκρινε τον κανονισμό και τη χρηματοδότησή τους μέσω του Connecting Europe. Το πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω σήμερα θα το μοιράσουμε εγώ και ο Ματθαίος Γκρός. Θα ήθελα να σας μιλήσω καταρχήν για τις μεταφορές και τις οικονομικές των επιπτώσεις. Να δούμε το TEN, να δούμε τα σχέδια υποβολής διαδρόμων, να δούμε τον απολογισμό των τεν και να δούμε τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε. Και αυτό ελπίζω να το κάνουμε γρήγορα για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Οι γενικότερες οικονομικές επιπτώσεις των μεταφορών. Η όλη πολιτική βασίζεται στην αρχή ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς με τις διασυνδέσεις που έχει αυτή με τον ευρύτερο κόσμο. Βράχοι και μεσοπρόθεσμες επενδύσεις κεφαλαίων στις μεταφορές μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ περισσότερη απασχόληση και ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα μπορούν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη οι έρευνες από την Κομισιόν και το Ινστιτούτο Φρανκόφερ καθώς και μία μελέτη που έχει προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις στην απασχόληση δεν είναι κάτι που το έχουμε ακόμη εξετάσει πλήρως αλλά για σήμερα να σας δώσω μόνο το ύψος γενικότερα των ε, κονδυλίων που αφορούν αυτά τα θέματα. Ήθελ, θέλησα να δω ποια θα ήταν η απώλεια, ποιο θα ήταν το κόστος της μη Ευρώπης. They suggested the total... Και ή λένε ότι οι συνολικές επενδύσεις από όλους τους διαδρόμους μέχρι το 13 30 θα ανέρχεται σε ύψος 622 δις. Επίσης φαίνεται ότι αυτού του είδους η δαπάνη θα δώσει ρυθμό ΑΕΠ πάνω από 5 προς 1. Και για, τις, για την απασχόληση 15 με 30 10 και μισό με 12 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Το άλλο σημείο που τονίζει η μελέτη είναι το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο των διαμεθοριακών συναλλαγών και μεταφορών ώστε να δημιουργηθούν καινούργιε αγορές που να εφαρμόζουν καινοτομία, πολιτικές καινοτομίας, μέσω των τέντι. Δεν έχω άλλες λεπτομέρειες, αλλά νόμισα ότι αυτοί οι γενικοί αριθμοί είναι ενδιαφέροντες. Τώρα τα TEN-T και το Connecting Europe. Όπως ξέρετε το Συμβούλιο και τα Κοινοβούλιο δέχτηκε το νέο πλαίσιο για τις υποδομές στα τέλη του 2013. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το τι θα έπρεπε να γίνει με τα κράτη-μέλη από εμάς ως συντονιστάς αναφέρονται από τον κανονισμό και οι δημοσιονομικές δυνατότητες μέσω του προπολογισμού και του Connecting Europe. Ο συνδυασμός αυτός κανονισμού και διαχείρισης χρηματοδότησης είναι κάτι βαθύτερο από οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα στα, για τα τέντη. Είναι μια προσπάθεια ποιοτικού άλματος από την κουρελού που υπήρχε προηγουμένως προς το πλήρες δίκτυο που θέλουμε να δημιουργηθεί. Για τον ίδιο τον κανονισμό, ο κάθε συντονιστής θα συντονίζει όλους τους τρόπους μεταφορών. Όχι πια δηλαδή έναν τρόπο αλλά όλους. Οδικές μεταφορές, σιδηροδρόμους, θαλάσσιες μεταφορές, ποτάμιες και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρόμων, RTMS. Εννέα διάδρομοι υπάρχουν μέχρι τώρα και ο χάρτης της Ευρώπης με τους διαδρόμους μοιάζει λιγάκι με το χάρτη του υπογείου του Λονδίνου με όλες τις διασυνδέσεις κλπ. Αυτοί οι νέοι διάδρομοι συμπληρώνονται και από τους λεγόμενους οριζόντιους διαδρόμους που πηγαίνουν παντού ο ένας αφορά και το ERTMS και ο άλλος τις θαλάσσιες μεταφορές. Ως συντονιστέ κάναμε πολλά. Όχι μόνο για να εξετάσουμε έναν έναν τους διαδρόμους, αλλά και συλλογικά όλους για να γίνουν αυτά που κάνουμε συνεπή σε όλες τις διαστάσεις τους. Και οι εννέα διάδρομοι και η γεωγραφική, και οι δύο οριζόντιοι τους διαχειρίζεται για το καθένα τους διαχειρίζεται ένα συντονιστής και πράγματι ο ρόλος τους είναι ένα από τα καινούργια στοιχεία στο καινούργιο σύστημα. Πέρυσι ο κάθε συντονιστής για τους εννέα διαδρόμους έχει υποβοηθηθεί και από εξωτερικούς συμβούλους. Πήραν τον κανονισμό και μέτρησαν ολόκληρο τον διάδρομο για κάθε τρόπο μεταφοράς ως προς τον κανονισμό για να δούνε πού υπάρχουν ελλείψεις, τι μεγέθους είναι οι ελλείψεις αυτές και πώς να λυθούν. Μα ζητήθηκε λοιπόν να δούμε ιδιαίτερα αν υπάρχουν χάσματα στις διαμεθοριακές επικοινωνίες και συγκοινωνίες γιατί φαίνεται ότι οι εταιρείες υποδομών και οι χώρες περιορίζονται στην επικράτειά τους η καθεμία και όχι και γύρω γύρω. Διαμεθοριακά λοιπόν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συνδυασμένες μεταφορές και interoperability. Αυτά είναι τα στοιχεία που θελήσαμε να εξετάσουμε. Συνεργαστήκαμε όλοι μαζί ως συντονιστές, ως κολέγιο συντονιστών. Και αν υπάρχει από τον κανονισμό ο διάδρομος, μία δομή διαχείρισης ε, και ένα σχέδιο εργασιών, που θα σας το εξηγήσω λίγο, τότε υπάρχει μια βάση για να γίνει έπια ποιότητα και υψηλές προσδοκίες. Και τμήμα είναι φυσικά, τμήμα τους είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία και στρέφουμε γι' αυτό στον Ματθαίο Γκρόσο. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενε πριν πάρει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πατ Κόξ ως πρόεδρος. Τώρα ο ματιού. Ε, μου ότι δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο. σε καλωσορίζω κι εγώ. Είχα την χαρά και την τιμή να είμαι μέλος τη Επιτροπή αυτής. Για πρώτη φορά στην ιστορία ε, στην τέταρτη φάση των διευρωπαϊκών δικτύων είναι η καινοτομία ότι έχουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο. Το 2013 συζητήθηκε αυτό και εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα όσα ανέφερε ο Πατ Κόξ. Και αν το δούμε και στην προετοιμασία των διαφόρων διαδρόμων, για μας τι έχει σημασία. Να πείσουμε τα κράτη-μέλη, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι τουλάχιστον το 80% του σιδηροδρόμου και της εσωτερικής ναυσιπλοείας ε, θα πρέπει να είναι το κέντρο βάρους και μέχρι ανανεώσιμες ενέργειες ε, αυτά δεν συνάδουν πάντα με κάποιες εθνικές προτεραιότητες όπως ξέρετε, διότι εμείς θέλουμε αυτό το δίκτυο. Διαπιστώσαμε επίσης γενικά στη χρηματοδότηση των ε, έργων ότι τα κέντρα βάρους που δίνουν και τις κατευθυντήριες γραμμές χρειάζονται μεγαλύτερη αποκέντρωση, επικουρικότητα. Και στο παρελθόν είχαμε λιγότερα χρήματα, αλλά ε, είχε σημασία η χρηματοδότηση. Ε, στο παρελθόν ήταν μέχρι 20%, τώρα είναι μέχρι 80% για τις χώρες συνοχής. Και για τις χώρες που δεν είναι συνοχή μπορεί να ε, έχουμε 40 με 50% επιδοτήσεις ή άμεση χρηματοδότηση. Αυτό είναι στοιχειώδες και στους δύο τομείς. Σε όλα τα έργα που έχουν υποβληθεί και έχουν συζητηθεί, η χρηματοδότηση είναι 30 με 40% αυτή που απαιτείται, δηλαδή για να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Και δεν μιλώ για τα μεγάλα, μπορεί να είναι και μικρότερα. Ε, ε ας πούμε στο σιδηρόδρομο υπάρχουν μικρά έργα για να κλείσουν κάποια παραθυράκια και κάποια ελλείμματα. Τώρα, απευθύνουμε την πρώτη έκκληση για την υποβολή έργων. Δεν μπορούμε να μπούμε σε όλε τις λεπτομέρειες τώρα. Όχι επειδή θέλουμε να σας κρύψουμε τίποτα, αλλά γιατί είναι στο στάδιο της ανάλυσης ακόμα. Είδαμε τα εξή δύο. 12 δισεκατομμύρια ευρώ ε, χρειάζεται από το Connecting Europe. Οι αιτήσει ε, υπερβαίνουν κατά πολύ τα 30 δις. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Αν δούμε τη σχέση των έργων ε, το συνολικό τους αθροισμά είναι πάνω από 120 δισεκατομμύρια. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που είπα προηγουμένως. Εάν θέλουμε να κλείσουμε κάποιες τρύπε, κάποια κενά, χρειάζεται 30 με 40% χρηματοδότηση. Και στην ανάθεση αυτών των έργων θα το διαπιστώσουμε. Και εκεί κινείται και όλη η συζήτηση που κάνουμε για το μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο στην Ευρώπη, όπου είμαστε πεπισμένοι ότι οι μεταφορές μπορεί να χρησιμοποιήσουν και αυτά τα μέσα, ανάλογα όμως με το μέσο μεταφοράς και τις υποδομές που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Θα πρέπει κάθε φορά να αναζητηθεί το σωστό εργαλείο, το χρηματοδοτικό, αναλόγως λοιπόν του μέσου και το τι θέλουμε να ενισχύσουμε. Ο συνάδελφος Μπόντεβικ ε, ο συνάδελφος έτσι έχουν κάνει μια πρόταση ε, που αναλύει τα διάφορα μέσα και τις δυνατότητες και ε, θα κάνουν και προτάσεις για τους διαδρόμους. Ανά κάθε διάδρομο ξεχωριστά θα μας πούν ότι για να φτάσουμε στον στόχο μας χρειάζονται τα εξής. ΣΔΙΤ καθόλου δεν αποκλείεται εκτός από την χρηματοδότηση και η μόχλευση και αυτή τη στιγμή Έχουμε και τα ομόλογα έργου ε, που είχαμε την ευκαιρία να το ψάξουμε αυτό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και διαπιστώσαμε ότι σε κάποιους τομείς το 10% που έχουμε και στη διευκόλυνση διασυνδέοντας στην Ευρώπη για τα χρηματοδοτικά μέσα ε, μπορούν να έχουν μια αμόχρευση μέχρι ε, της τάξης του 30. Δηλαδή δεν αποκλείεται καθόλου αυτό, απλώς θα πρέπει να βρει τη σωστή επένδυση που εφαρμόζεται κάθε φορά. Περισσότερο στις λιμενικές υπηρεσίες και στις ε, υποδομές για τους αυτοκινητοδρόμους και τις πλατφόρμες εφοδιαστικής. Εκεί περισσότερο υπάρχει μόχλευση. Ε, έχουμε το πρόγραμμα εργασίας, ε, Σε τέλη του έτους το καταθέσαμε. Συζητήσαμε βεβαίως κατευθυντήριες γραμμές με τα κράτη-μέλη και έχουμε συνεννοηθεί για την προετοιμασία μας μαζί τους. Αποτέλεσμα, ε, ε, έχουμε μια ανάλυση αναδιάδρομο, τα είπε και ο Σάφος με στοιχεία υποδομής, κοινωνικά, ε, οικονομικά, περιβαλλοντικά, ας πούμε εσωτερική ναυσιπλοεία σε ορισμένες περιοχές. Είναι πολύ προβληματική, δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάσει οικολογία με οικονομία στα πλωτά ποτάμια και περιμένουμε τις προτάσεις, όλες οι προτάσεις έγιναν δεκτές από όλα τα κράτη μέλη, αλλά είμαστε ακόμα ε, στη διαδικασία που, η οποία τρέχει και αναμένεται να ολοκληρωθεί ε, στα τέλη του εξαμήνου. Ε, βελτιώνουμε τώρα τις δυνατότητες με αυτή την περίφημη ανάλυση του Ινστιτούτου Φράουενχόφερ που αναλύει και τα κοινωνικά και τα οικονομικά στοιχεία ας πούμε, δημιουργία θέσεων εργασίας και αυτά τα αναλύουν. Και η μελέτη αυτή ε, ε, προσέχει περισσότερο και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν θέλω να μεταφέρω ε, τις μεταφορές από τον αυτοκινητόδρομο στο σιδηρόδρομο σε ένα διάδρομο, τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Γιατί πολύ συχνά αυτά τα στοιχεία δεν λαμβάνονται ε, επαρκώς υπόψη όταν γίνεται οικονομική ανάλυση ενός έργου. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Πατ Κόξ ε, για τον απολογισμό του πρώτου έτους. Ε, εγώ είμαι πολύ καινούριο, θα τα πει ο συνάδελφος Πατ Κόξ αυτά, για την ανάλυση του πρώτου έτους λειτουργίας αυτού του Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη όλα τα, όλους τους γεωγραφικούς ε, διαδρόμους έτσι ώστε να μπορέσουν να εμπλακούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Προσπαθούμε ε, να τους προσεγγίσουμε γιατί δεν μπορούν να γίνουν αυτά σε μία μέρα. Επίσης έχουμε την βοήθεια των συμβούλων που είδαν τον κανονισμό και μας είπαν που υπήρχαν ελλείψεις και πώς μπορούμε να ορίσουμε τις προτεραιότητες. Επίσης, ο καθένας για τους γεωγραφικούς διαδρόμους έπρεπε να υποβάλει ένα γραπτό σχέδιο εργασίας που υποβάλαμε στα κράτη-μέλη, στα εμπλεκόμενα κρατη ε, αυτά τα προγράμματα εργασίας έχουν εγκριθεί κατά μείζωνα λόγο. Είδαμε ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά θα δοθεί τελική μορφή όταν φτάσουμε στον τελικό απολογισμό σε μερικές εβδομάδες. Λάβαμε είχαμε πολύ θετική και εκτενή συνεργασία από τα κράτη της περιφέρειας, τους ε, διαχειριστές και ούτω καθεξής. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μοντέλο συνειδιοκτησίας διαδρόμων και έτσι έχουμε μία πολύ καλή βάση για μελλοντικές εργασίες γιατί δεν επιβάλαμε ένα πρότυπο σε άλλους, υπήρξε μία συνεργασία άρα υπήρχε μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και τούμπαλιν. Επίσης οι συντονιστές ε, συνεργάστηκαν για να υπάρχει συνέπεια, συνεκτικότητα και για να μπορέσουμε να αποστείλουμε ε, ένα εκτενές και συνεκτικό μήνυμα. Στο Μιλάνο είχαμε ένα άτυπο συμβούλιο υπό Ιταλική Προεδρία και έχουμε ομάδες συντονιστών που επισκέπτονται τις πρωτεύουσες όπου υπάρχει διασταύρωση διαδρόμων και το είδαμε στην Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία σε τη συνεργασία σε υπουργικό επίπεδο για να δούμε και τι επενδύσεις μπορούν να γίνουν. Κατά την περίοδο συνεργασίας το σχέδιο Juncker και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είδε το φως και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι διοχετεύονται ορισμένα χρήματα εκεί και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κινητοποιηθούμε για να φτάσουμε στη κινητοποίηση μέσω των διαδρόμων. Και αυτό θα το προωθήσουμε όπως είπαν και οι συνάδελφοι Μποντεβίκ και Σέκη. Επίσης είχαμε στο Ίνσπρουκ μία διάσκεψη όπου είδαμε τα βασικά προγράμματα μέσω διαδρόμων έτσι ώστε να προβαίνουμε σε μία κοινή εργασία. Δηλαδή ε, είναι ένα μέσο διασταύρωση στοιχείων ως προς τους διασταυρούμενους αυτούς διαδρόμους και όπως σας είπα μας ενδιαφέρουν οι διασυνοριακές στενοποί και οι συνδυασμένες μεταφορές. Δεχόμαστε όμως ότι τον πρώτο χρόνο ένα μεγάλο μέρος της εργασίας μας αφορά τις παραδοσιακές ελλείψεις υποδομών και θα πρέπει να δούμε το πρασίνισμα των διαδρόμων, τα ευφύ συστήματα διαχείρισης, τα βιώσιμα δίκτυα αστικών ή υπεραστικών μεταφορών και όλες τις προκλήσεις οι οποίες θα μας φτάσουν σε μια στρωματοποίηση, στρωματοποίηση της κατανόησης του όλου ζητήματος. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να το δούμε σε επίπεδο ε, βιομηχανιών, υπηρεσιών, στα πλαίσια της ψηφιοποίησης, των ε, εναλλακτικών καυσίμων για τα λεωφορεία και ούτω καθεξής. Τέλος, προσβλέποντας σε μία μελλοντική ανάπτυξη, θα ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς θα συμμετάσχετε στους ε, διαλόγους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών σας τα προγράμματα εργασίας θα αναθεωρηθούν το 16 και κάθε δύο χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε ορισμένους τομείς όπου ε, είχαμε επιταχύνσεις ενώ αλλού είχαμε επιβράδυνση. Θέλουμε λοιπόν να κινηθούμε δυναμικά και αυτή θα είναι και η μελλοντική πορεία των σχεδίων μας. also zum Abschluss ganz kurz Πολύ σύντομα, τα χρήματα και τα κονδύλια που έχουμε ε, τώρα στη διάθεσή μας θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με φιδό. Ακούσαμε για 500 δις ε, επενδύσεις. Ξέρετε τι είναι το Connecting Europe και ποια μέσα έχει, αν το δούμε και με τη μόχλευση και με αισιοδοξία μπορούμε να πούμε 210 μέχρι 220 ε, δις αυτή την πενταετία μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αρχή, αλλά σε καμία περίπτωση το δίκτυο που φιλοδοξούμε να έχουμε μέχρι το 2030 ε, στην πλήρη του και έτοιμη μορφή. Το δεύτερο σημαντικό για μένα στοιχείο και για τους υπόλοιπους συντονιστές. Η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, να ζητούμε και επιζητούμε την επαφή με τις περιφέρειες, τους δήμους και κοινότητες και τις ε, διάφορες οργανώσεις περιβαλλοντικές και άλλες ΜΚΟ, έτσι για να υπάρχει μια διαβούλευση, ένας διάλογος στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και όχι αργότερα με άλλες μορφές. Εμείς είμαστε και παραμένουμε πεπισμένοι ότι για να κερδίσουμε τους πολίτες στο πλευρό μας θα πρέπει να είναι πολύ σωστά ενημερωμένοι σε βάθος και εκτενέστατα τα επόμενα χρόνια αυτό θα είναι μεγάλη προτεραιότητα. Για την κινητικότητα, για τις μεταφορές έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, έχουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο, έχουμε πρόγραμμα εργασίας, έχουμε συνολική ανάλυση όλων των χρηματοδοτικών μέσων, έχουμε ανάλυση επιπτώσεων και αντικτύπου σε περιβάλλον, οικονομία και εργασία, απασχόληση. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι σε συνεργασία μαζί σας να προωθήσουμε ε, αυτή την υπόθεση και με χαρά θα μοιραστούμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ και τους δύο για την εισαγωγή σας και τώρα έχουν το λόγο οι δικοί μας συντονιστές. Πρώτος ο Βίμ Παντενκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή να υποδεχόμαστε εδώ τους κυρίους Κόξ και Γκρός είναι κορυφαίοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην βουλευτές, και υποθέτω ότι όλα αυτά που μάθανε εδώ τα χρησιμοποιούν και τα εφαρμόζουν στη σημερινή τους δουλειά ως συντονιστές. Και πραγματικά μπορούμε να αναμένουμε πολλά και από τους δύο. Και δεν μιλώ εδώ για τεχνάσματα, αλλά για δεξιοτεχνία. Ε, αυτό που θέλω να πω τώρα, φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι τα οικονομικά. Ο κύριος Κόξ αναφέρθηκε λίγο σε αυτό και ο Ματιό Γκρός. Τώρα βρισκόμαστε στη διαβόλευση την ε, κοινοβουλευτική του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και ως Επιτροπή Μεταφορών ε, χρειάστηκε να καταπιούμε το γεγονός ότι έχουν πάρει λεφτά από το Connecting Europe στην ενδιάμεση έκθεση του κυρίου Κριστόφερσον θα μπορούσατε να δείτε σαν προέκταση αυτής μια εναλλακτική δυνατότητα χρηματοδότησης. Κάπου αυτό αναφέρεται, αλλά έτσι ακροθυγός. Υπάρχει περιθώριο, μπορεί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να είναι ενίσχυση ή μπορούμε να έχουμε μεικτή χρηματοδότηση, ΣΔΙΤ, ΣΕΦ, ιδιώτες, ΣΕΦ, crowdfunding, ε, ΣΕΦ, ε, ΕΦΣΥ, θέλω να με ενημερώσετε. Μετά, ποια είναι η σχέση μεταξύ του βασικού δικτύου και του συνολικού δικτύου, αυτό το comprehensive. Τι σημαίνει αυτό, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, γιατί μας ρωτούν πάρα πολλοί πολίτες εκτός από το βασικό ε, δίκτυο, όλες αυτές οι ερωτήσεις ανήκουν στο γενικότερο, όχι στο βασικό. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, ε, το έχετε υπόψη σας και στο μυαλό σας ξεκάθαρα. Συμφωνώ με τους δύο κυρίους, είναι από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα αυτή τη στιγμή και έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει ε, να παραμείνουμε σε αυτό όμως και να μην επεκταθούμε. Για την, ε, τις τώρα. Ε, λέει ο κύριος Κόξ ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Ωραία. Αλλά αν δούμε πώς γίνεται αυτή τη στιγμή η αδειοδότηση και η έγκριση στην Ευρώπη και εδώ σέβομαι απολύτως ό,τι θέλετε και τη βιωσιμότητα και τη διαβούλευση αλλά τώρα ε, ε, στη Γερμανία προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη γραμμή Betue που ξεκινάει από την Ολλανδία και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις. Μπορείτε αυτό να το επιταχύνετε. Και επίση τι γίνεται με τον οριζόντιο συντονιστή, ε, τον κύριο Σίμψον, για τις λεγόμενε θαλάσσιες λεωφόρους. Αυτός συμμετέχει αρκετά επαρκώς ε, στις περιφερειακές, ε, πώς να το πω, στους γεωγραφικούς διαδρόμους, όχι τους θαλάσσιους. Δηλαδή μόνο με τη θάλασσα ασχολείται ο κύριο Σίμψον. Αλλά συνδέεται αυτό και με τους υπόλοιπους εννέα διαδρόμους. Και μια ερώτηση για τη χρηματοδότηση από τις χώρες συνοχής. οι οποίες είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μέσα TNT. Ε, για τα λιμάνια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια από τη συνοχή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι χώρες ε, αυτές δεν θέλουν από τα κονδύλια των διευρωπαϊκών δικτύων να χρηματοδοτήσουν λιμάνια, αλλά απαλού. Γιατί τα θέλουν για τους δικούς τους λόγους. Και τώρα η αλλαγή τρόπου μεταφοράς, αυτό το περίφημο ε, modal shift, δική σας ιδέα ήταν αυτή κύριε Γκρός, δική σας η λευκή βίβλος και τώρα είμαστε στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, γίνεται λόγος για συνδυασμένες μεταφορές, co-modality το λένε αυτό. Άλλο το modal shift που είναι η, μετακίνηση, η μετατόπιση από τον ένα τρόπο μεταφορά στον άλλον. Ε, είναι κάπως επιτακτικό αυτό και το θέμα είναι αν θα το επιλέξει η αγορά. Και μετά για τη συντήρηση. Ε, τα τελευταία χρόνια, ή το τελευταίο έτος τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάμε πάρα πολύ για τη συντήρηση. Ε, δεν θέλουμε κάθε φορά να φτιάχνουμε νέους αυτοκινητοδρόμους, καινούργια έργα υποδομής. Συνήθως η προτεραιότητα είναι η συντήρηση των υφισταμένων υποδομών και δικτύων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ εξ ονόματος της δικής μου ομάδας να καλωσορίσω τον συνάδελφο Γκρός και Κόξ και να τους ευχαριστήσω για τα όσα μας παρουσίασαν. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ως εξή. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει ακόμα είναι, τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα, ότι για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω σίγουρα της νέας δομής των διευρωπαϊκών δικτύων έχουμε συνεργασία των συντονιστών των δικτύων για πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντικό να μην προσπαθεί ο κάθε συντονιστής να κάνει τα δικά του στο δικό του δίκτυο αλλά πραγματικά να υπάρχει ανταλλαγή και συνεργασία μεταξύ ε, των εννέα συντονιστών σε αυτή την ομίγυρη εκεί. Ε, πάρα πολύ σημαντικό γιατί και αυτό ε, θα φέρει συνέργειες και προστιθέμενη αξία. Άλλο θετικό που σημείωσα είναι το εξής. Και είναι και το μοναδικό έτσι και στη σημερινή δομή. Αυτό το είπατε εσείς κύριε Κόξ, learning by doing μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια δηλαδή της υλοποίησης. Ε, τα Υπουργεία Συγκοινωνιών και Μεταφορών δεν διακρίνονται για τη φιλοευρωπαϊκή του τάση, το λέω έτσι ε, προσεκτικά ε, και συγκρατημένα. Προσπαθούμε αυτούς τους κυρίους εκεί που στα Υπουργεία είχαν πολύ εθνοκεντρική στάση, να τους μάθουμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες και άλλες λύσεις που μπορεί να είναι και καλές και μπορούμε να διδαχθούμε από τους άλλους και να έχουμε συνέργεια και συνεργασία. Γενικά λοιπόν... Ήταν από τα καλύτερα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα δηλαδή τα τελευταία χρόνια από τις καλύτερες ιδέες ε, ε, με βεβαίω ε, στο πλευρό τους πάντα δραστήρια και ενεργή υποστήριξη των δύο συνομοθετών, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προήλθε αυτή η πρωτοβουλία. Ε, θέλω να κάνω και ερώτηση και παρακαλώ να μου την απαντήσετε αν μπορείτε. Ο συνάδελφος Γκρός μου έκανε εντύπωση ότι είπε ότι τα προγράμματα εργασίας θα έχετε συνεννοηθεί με τα κράτη-μέλη και ο κύριος Κόξ προσέθεσε στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Υπάρχουν κράτη-μέλη που, ε, που είναι υποδειγματικά στη συνεργασία τους και κάποια άλλα που είναι κάπως διστακτικά, που χρειάζονται λίγη μεγαλύτερη υποστήριξη για να προχωρήσουν. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Ερώτηση δεύτερη. Στην έκθεσή σας διαπίστωσα ότι λόγω των δυσκολιών που είχαμε στο παρελθόν με το RTMS στο σιδηρόδρομο, τώρα σκέφτεστε λέει ένα πρόγραμμα RTMS Breakthrough, ένα ρηξικέλευθο πρώτη. Αυτά είναι πολύ μεγαλόστομα. Τι ακριβώς εννοείται και τι, σε τι αποσκοπείτε. Δεν κατάλαβα απολύτως. Τρίτη ερώτηση. Μας στείλατε κάποια έγγραφα, είχατε την καλοσύνη και εκεί αναφέρεται και το εξής. Κάθε πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εκτίμηση που βρίσκεται το κάθε κράτος μέλος απέναντι στα υπόλοιπα για τη διαλειτουργικότητα ε, και τις συνδυασμένες με τα διατροπικότητα όπως λέγεται. Αυτό πότε θα το έχετε στα χέρια σας και πότε θα μας το στείλετε και εμάς. Και η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, γιατί είναι σαφές νομίζω αυτό το σημείο, το μήνυμα, ότι θα ότι έχετε ε, προκηρύξει έργα για 12 δισεκατομμύρια και σας ήρθαν προτάσεις για 30 ε, και ενδιαφέρον. Οπότε, επειδή ήμουν και συγητής, ε, στην περασμένη περίοδο, την περασμένη θητεία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ήξερα πόσο δύσκολο ήταν να ε, επιβληθούν τα ομόλογα έργου απέναντι και στα κράτη-μέλη. Και θέλω να ρωτήσω, τα ομόλογα έργου τα συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν το παρακολούθησα καλά και αν το θυμάμαι καλά, έχουμε 250 εκατομμύρια τότε ε, πιλωτικά απελευθερώσει και έκτοτε συγγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είχε αυτό ε, απόδοση, ε, τι συνέχεια δόθηκε, ήταν θετική, ήταν αρνητική, χάθηκαν. Ε, αν δεν απέδωσαν όσο θα επιθυμούσαμε, δεν χάλασε και ο κόσμος, αλλά να μάθουμε τι έγινε. Και κάτι άλλο που είναι επίσης μοναδικό και καθόλου εύκολο να το επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη ήταν η συμμετοχή ε, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και το είπαν και οι δύο συνάδελφοι σήμερα, αν δεν συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες δεν θα ε, καταστεί δυνατό τέτοια μεγάλα έργα να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 20 και 30 χρόνια. Αν το παρακολούθησα καλά, υπάρχουν διαφορετικές ε, μέθοδοι στα διάφορα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη είναι αρκετά άκαμπτα όταν μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα των διαδρόμων και υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που είναι λίγο πιο ανοιχτά και φιλελεύθερα και ευέλικτα. Οπότε ρωτώ, τι εμπειρίες έχετε με τα διάφορα κράτη-μέλη και πώς σας φέρθηκαν. Ευχαριστώ. Η Τζάκι Φώστερ. Πίτερ Φαντάλ. Ο Πίτερ Φαντάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, στην πολιτική συχνά γίνεται λόγος για το εφικτό. Πώς μπορεί η πολιτική να διαμορφώσει μια εφικτή κοινωνία, να αλλάξει τον κόσμο. Ε, συχνά αυτό δεν το καταφέρνουμε, αλλά εδώ ε, ε, στη συγκεκριμένη πρόταση είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να αλλάξει την κοινωνία μας. Ε, τις υποδομές με τους διαδρόμους, τις διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Είναι κάτι που πραγματικά μπορούμε να επιτύχουμε, να αλλάξουμε τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω λοιπόν εγώ τις εξής δύο ερωτήσεις. Πρώτον, τα οικονομικά. Για τη δική μου πολιτική ομάδα ήταν τεράστια απογοήτευση αυτά που πρότεινε ο κύριος Γιούνκερ για το επενδυτικό του σχέδιο. Γιατί έκανε όλες αυτές τις ωραίες δηλώσεις και μετά πήγε και πήρε τα λεφτά από το Connecting Europe και τα TNT. Ε, τι μας λένε οι δύο κύριοι ε, μήπως είμαστε εμείς ιδιαίτερα απεσιόδοξοι, εσείς είστε αισιόδοξοι, ελπίζετε ότι ε, μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το σχέδιο Juncker προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερη ερώτηση. Για ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο συγκεκριμένο, ε, πολύ συχνά το βρίσκουμε αυτό στα έργα υποδομών. Είναι η περίφημη ανάλυση κόστους ωφέλειας. Όταν κάνεις ένα έργο ε, υποδομών, πάντα γίνεται μια τέτοια ανάλυση, έτσι, κόστους κόστος-οφέλους. Και ε, διάφορα προγράμματα δεν επιλέγονται ε, διότι θεωρείται ότι η ωφέλεια που θα προκύψει σε σχέση με το κόστος είναι πολύ μικρή. Και ένα από τα στοιχεία που λαμβάνεται υπόψη είναι η χρόνια απόσβεσης. Αυτό αφορά και διάφορα κανάλια στην εσωτερική ναυσιπλοεία που είναι 25 χρόνια συνήθως η απόσβεση. Αυτό πρόεδρε το θεωρώ παράλογο. Αν δείτε ε, ότι ε, αν είναι αυτοί 25 χρόνια δεν πρόκειται να κατασκευαστεί κανένα κανάλι, ε, καμία τέτοια εσωτερική πλωτή, τεχνητή πλωτή οδός, διότι δεν είναι 25 χρόνια η απόσβεση, είναι πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό το έχετε σκεφτεί γιατί τόσο μικρή, τόσο σύντομη περίοδος για τέτοια έργα που καμιά φορά αποδίδουν μετά από 100 χρόνια δεν είναι εφικτή. Αυτά πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο συντονιστές για την έκθεσή του και τον Πατ Κόξ και τον Ματιό Γκρός, πρώην συνάδελφο εδώ στην Επιτροπή μας. πολλά υπόθηκαν, θα κάνω ερωτήσεις, ε, αλλά να πω κι εγώ κάτι εισαγωγικά. Ήμουνα και εδώ και την περασμένη θητεία και έχω την αίσθηση ότι αυτό το TNT που στο χάρτη είναι σαν χάρτης ε, του μετρό του Λονδίνου και για μένα από τότε που είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο αγαπημένος μου χάρτης γιατί φαίνεται ότι έτσι μπορούμε να συνδέσουμε την Ευρώπη και είναι σαν ένα μετρό. Ωραία όλα αυτά λοιπόν, το ΣΕΦ, Connect Europe, το TNT ήταν πολύ μεγάλο επίβολο σχέδιο. Ακόμα και αν δεν πήραμε τα χρήματα που επιθυμούσαμε είναι τριπλάσια από τα προηγούμενα. Και ε, γι' αυτό και οι συντονιστές είναι για μας οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Έτσι σας βλέπω γιατί όλοι όσοι θέλουμε να εφαρμοστούν αυτά τα έργα θέλουμε να πιάσουν και τόπο τα λεφτά. Υποθέτω λοιπόν ότι εσείς θα πείτε ως συντονιστές, δεν ξέρω αν θα το πείτε δεν θα το πείτε, σας το λέω εγώ. Ε, όταν ο κύριος Γιούνκερ ας πούμε θέλει να κάνει το ταμείο του να του πείτε να μην τα πάρει τα λεφτά από το Connecting Europe. Ερωτώ, το είπατε αυτό και θα γνωρίζετε και τις προτάσεις ε, του σχεδίου Juncker για τις μεταφορές, οι οποίες ε, αφορούν και τους δικούς σας διαδρόμους. Βέβαια είναι περισσότερο αυτοκινητόδρομοι και λιγότερο σιδηρόδρομοι και εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, δεν είναι πάρα πολύ στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών, αλλά πώς το αξιολογείτε και επίσης σας ρώτησαν καθόλου για να τα προτείνουν αυτά. Και μια ερώτηση προς τον Πατ Κόξ. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη ε, συνήθως τα περισσότερα ε, είναι συνεργάσιμα. Και θέλω να ρωτήσω, όπως ρώτησε και ο Ισμαήλ Ερτούκ, ε, ποια δεν είναι συνεργάσιμα ή διστάζουν ένα πρόθυμα, για να πάμε οι βουλευτές να πιέσουμε λίγο τις χώρες μας. Έχω την αίσθηση ότι καμιά φορά η Γερμανία έχει ανάγκη λίγο υποστήριξης έτσι, και όθησης. Κύριε Κόξ, έχετε ε, στο δίκτυό σας ένα σημείο που έχει προβλήματα. Ε, ε, είναι μια διασύνδεση Βερολίνο-Κίελο και ρίχνει ο ένας το μουτζούρι στον άλλον, τον μπαλάκι. γιατί υπάρχει ένα προβληματικό σημείο στο Φίμερ Ζούντ και Φίμερ Βέλτ είναι στενοπός ε, και θα δημιουργηθούν εμποτιλιαρίσματα εκεί ε, στο έργο αν δεν λυθεί αυτό το, θέμα στο συγκεκριμένο διάδρομο. Και ε, να ρωτήσω το Ματιό Γκρός, είπες για την εσωτερική ναυσιπλοεία ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την οικονομία με την οικολογία που δεν είναι πάντα πράγμα εύκολο. Τι εννοείς ακριβώς, νομίζω ότι κατάλαβα, αλλά μπορείς να μας πεις αφορά ποια ποτάμια τον Έλβα, στην διεύρυνση ποταμών της Κίτης. Ε, επίσης είπες ότι έρχεται επαφές με περιβαλλοντικές οργανώσεις, επί τόπου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν μεγάλα έργα υποδομών, συγκοινωνιών, μεταφορών που είναι πολύ σημαντικά και ε, να βαγούν εκεί, ε, γιατί δεν έχουν συνεννοηθεί με τους πολίτες. Στη Γερμανία είναι έργο που ονομάζεται Επιτροπή Υψηλών, 20 χρόνια σχεδίαζαν, Ανόβερο, Αμβούργο, Βρέμι ήταν μια σιδηροδρομική σύνδεση αυτή που δεν είδε ποτέ το φως ε, και ε, δεν ευδοκίμησε πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ η Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συντονιστές, σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας και καλή τύχη για τη συνέχεια. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πείτε ποιο όραμα έχετε για το μέλλον της χρηματοδότησης των δικτύων αυτών στην Ευρώπη των TNT. Τι καινούργια σχέδια υπάρχουν μετά από τη δημιουργία του επενδυτικού ταμείου. Θεωρείτε ότι αυτό το νέο ταμείο θα μπορέσει να μονιμοποιηθεί με όλες τις, με ό,τι σημαίνει αυτό και πώς βλέπετε την ψηφιοποίηση των μεταφορών και γενικότερα της χρήσης των λεγόμενων έξυπνων εργαλείων στις μεταφορές. Θα είναι κάτι καλό αυτό ή απειλητικό σε σύγκριση με αυτό που έχουμε τώρα, το RTT θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αλλά εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τις υπάρχουσες δυνατότητες και την τεχνογνωσία που έχουμε για αυτά τα συστήματα. Μήπως αυτό μειώσει τις ανάγκες μας και δεν χρειάζεται πια τόσο πολύ χρήμα για τη δημιουργία υποδομών τέτοιας έκτασης ή μεγέθους. Μήπως θα υπάρχει μικρότερη ανάγκη για μετακινήσεις με ατομικό ιδίως όχημα, περισσότερες συγκοινωνίες μαζικές και μήπως επίσης δεν χρειάζεται και τόση χρηματοδότηση πια. Θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών που να χρησιμοποιεί όλη την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μέχρι τώρα ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας ολόκληρη την κοινωνία. Εσείς οι συντονιστές πώς το βλέπετε αυτό. Υπάρχουν ακόμη φραγμοί για την ανάπτυξη των δικτύων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές. Κύριε Γκρός, είπατε κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Είπατε ότι θα δώσουμε οικολογικό χαρακτήρα στους διαδρόμους. Επειδή ανήκω στο κόμμα των οικολόγων, θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό τον οικολογικό χαρακτήρα που θα προσδώσετε στους διαδρόμους. Είπατε κάτι το οποίο αληθεύει. Ήσασταν ευρωβουλευτής. Εγώ δεν σας γνώριζα τότε. Αλλά στην παρουσίασή σας είπατε κάτι που με εξέπληξε. Είπατε ότι εσείς ως Ευρωβουλευτές, εμείς δηλαδή, ότι ο ρόλος μας, η αποστολή μας είναι να εκπροσωπήσουμε αυτές τις ε, νέες υποδομές. Να είμαστε οι πρεσβευτές αυτών των νέων υποδομών. Αλλά μπορείτε σήμερα να μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο εσείς θα βοηθήσετε τους ευρωβουλευτές, τους εκπροσώπους των πολιτών να συμμετάσχουν, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εμείς πρεσβευτές, εάν εσείς τη μεθοδολογία δεν συμπεριλαμβάνετε και τους ε, κατοίκους, διότι ίσως οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών να μην ε, είναι υπέρ συγκεκριμένων προγραμμάτων και σχεδίων. Τώρα, πώς η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας των Σιδηροδρομικών Δικτύων, πώς ε, εμπλέκεται με τους ε, διαδρόμους, ε, γιατί μιλάμε και για το τροχαίο υλικό και για την υποδομή γενικότερα. Και μία άλλη ερώτηση και προς τους δύο. Πώς θα συντονίσετε τα δίκτυα διαδρόμων με το ε, σύστημα των διατροπικών μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορών. Πώς το προβλέπετε αυτό. Ευχαριστώ Πέτερ Λούτκρεν. Okay, ε, Dann kommt Luis de Grandes Pascal. Καλά, τότε ο Luis de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να καλωσορίσω και τον κύριο Κόξ και τον κύριο Γκρός. Εγώ σας γνωρίζω σε αντίθεση με την προλαλή σας. Ε, ο κύριος Γκρός γνωρίζει πολύ καλά και τα θετικά και τα αρνητικά μας, ε, γιατί προέρχεται από μια συγκεκριμένη περιοχή. Μιλήσατε για πρεσβευτές αυτών των σχεδίων και προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την Ισπανία, αλλά ίσως είναι και γενικότερα. Γιατί πώς ε, εμείς σαν πρεσβευτές μπορούμε να επηρεάσουμε για να λυθούν αυτές οι διαφορές εκεί που υπάρχουν στους διαδρόμους. Εμείς έχουμε δύο διαδρόμους του Ατλαντικού και του, της Μεσογείου. Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα με τη Γαλλία διασυνοριακά. Πολλές φορές ευθύνεται η Γαλλία, άλλες φορές ευθύνεται η Ισπανία και αυτό αφορά και την ε, Πορτογαλία, διότι έχουμε προβλήματα ως προς μία πολιτική διάσταση των ε, ζητημάτων. Η Πορτογαλία ε, δεν θέλησε να προωθήσει το θέμα του, των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας των ΑΒΕ για λόγους καθαρά οικονομικούς. Αυτό είναι νόμιμο και δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει πάντα η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Υπάρχουν προβλήματα πολλές φορές για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα συνοριακά καθαρά προβλήματα, τα διασυνοριακά. Πώς μπορούμε εμείς ως πρεσβευτές να το αντιμετωπίσουμε το θέμα, διότι υπάρχουν δυσκολίες ε, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες, ιδιαίτερα σε διασυνοριακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ και δεν ξέρω κατά πόσο ε, ε, μπορούμε να, πούμε ότι σας γνωρίσουμε όλοι όλους. Τον κύριο Κόξ τον γνωρίζω πολύ καλά και αυτό που, μας, ε, που με ενδιαφέρει είναι ο διάδρομος της δικής μου περιφέρειας. Με ενδιαφέρει και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων γιατί ε, όταν ορίστηκε ένα από τα προγράμματα δεν υπήρχε το συνδέοντα στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, ε, δεν υπήρχε λοιπόν το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων όταν πρωτοϋποβλήθηκαν αυτά τα σχέδια. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα χάσματα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ως προς τον προγραμματισμό. Μπορείτε να, ε, μπορούν να εμπλακούν περισσότερα σχέδια και πώς μπορούμε να συνδέσουμε σχέδια, άρα μικρότερα, άρα μεγαλύτερα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το bundling και πώς μπορεί να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην χρηματοδότηση αυτή. Ντομινίκ Κρικέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ματιέ Γκρός και ο Πατκόξ είναι πολύ γνωστοί συνάδελφοι και θα ήθελα να τονίσω ότι και η ίδια η ύπαρξη των συντονιστών των διαδρόμων μας είχε ενδιαφέρει πολύ και μας και την Κομισιόν όταν συζητούσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για το Connecting Europe. Και τώρα τρέφεται το ένα πρόγραμμα από το άλλο. Ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι και να θέσω και ένα δύο ερωτήματα. Καταρχήν μία δημοσιονομική χρηματοδοτική δήλωση, διότι οι επενδύσεις στους διαδρόμους υπόκεινται στην δημοσιονομική δυνατότητα. Έκανα έναν υπολογισμό ενδιαφέροντα ως προς το Connecting Europe όπου θέλουν να περικόψουν ορισμένα κονδύλια του. 50 δισεκατομμύρια διέθετε στην αρχή, επί των οποίων τα 30 για τις μεταφορές, 10 για την ενέργεια και 10 για τις τηλεπικοινωνίες. Τα 30 λοιπόν δισεκατομμύρια των μεταφορών μεταφράστηκαν σε 23 μετά τις περικοπές του Συμβουλίου, το οποίο πάντοτε περικόπτει. Τελικά όμως έγιναν 13, διότι 10 δισεκατομμύρια προέρχονταν από το Ταμείο Συνοχής και απλώς είχαν ετικετοποιηθεί για αυτή τη θέση. Δεν ήταν πρόσθετα κονδύλια για τις μεταφορές, απλώς μεταφέρθηκαν από το κεφάλαιο 2 στο κεφάλαιο 1. Μένουν λοιπόν 13 εκατομμύρια για την ανταγωνιστικότητα και τις μεταφορές από το Connecting Europe. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν που τη στηρίζει και το Συμβούλιο είναι 2,7 δισεκατομμύρια από αυτά τα 13 να τα πάρουν για το σχέδιο Juncker. Άρα κατεβαίνουμε στα 10,3 δισεκατομμύρια. Και σκέφτηκα ότι 10,3 δις είναι ακριβώς το ποσό που είχαμε διαθέσει και στα προηγούμενα πολυετή σχέδια του προϋπολογισμού για, για τη δραστηριότητα της υπηρεσίας για τα μεγάλα δίκτυα. 8 δισεκατομμύρια ήταν πριν από 10 χρόνια και μετά μεταφράστηκαν σε 10,3 που είναι το μόνο που μένει πια από το Connecting Europe το οποίο είναι σαν να έχει εξαφανιστεί δημοσιονομικά. Δεν έχει πια λεφτά. Επανήλθαμε στην πρόταση προδεκαετίας της Κομισιόν να χρηματοδοτήσει κατά 8 δισεκατομμύρια αυτή την υπηρεσία δηλαδή. Θα το θυμούνται ορισμένοι. Επομένως πρέπει να ξέρουμε ότι το Connecting Europe εξαφανίζεται δημοσιονομικά από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Δεύτερον, αυτό που είπε ο Ισμαήλ. Τα ομόλογα έργου, σύμφωνα με τον κανονισμό του Γιούνκερ, είναι ακριβώς ο μηχανισμός των ομολόγων έργου, δηλαδή μια εγγύηση κινδύνου. Η πρώτη ανάληψη κινδύνου μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, equity ε, διάφορα άλλα τέτοια. Στην πράξη όμως το εκπληκτικό είναι ότι τα κράτη-μέλη είχαν ταχθεί κατά των ομολόγων έργου για το Connecting Europe και τώρα τα δέχονται, δέχονται με ενθουσιασμό για το σχέδιο Juncker για να εγγυηθεί τις απώλειες. Είχαμε μιλήσει για 250 εκατομμύρια για τα ομόλογα έργου, ένα είδος μικροσχεδίου Juncker δηλαδή, και ενεκρίθησαν 8 σχέδια κανένα από τα οποία δεν ανταποκρίνεται σε υποδομές μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι για πολλά σχέδια, όχι μάλλον όλα, δεν υπάρχει σύνδεση. Και θα ρωτήσω τους σύνδεση μεταξύ σχεδίων μεταφορών και του σχεδίου Γιούνκερ. Δηλαδή να μην αναμένουμε ότι οι εγγυήσεις δανείων ή για τις πρώτες απώλειες θα λειτουργήσουν έτσι. Απλό λοιπόν το ερώτημά μου. Οι συντονιστές μήπως μπορούν να μας κάνουν κάποια εκτίμηση για το σύνολο των σχεδίων για τα 615 δισεκατομμύρια που ανέφερε ο Πατ Κόξ. Πόσα από αυτά τα σχέδια θα έχουν κάποιο κέρδος 20%, 30%, 50%, 80% ή ακόμα λιγότερα. Ευχαριστώ πολύ. Η Σάσκουν Μπιλμπάου. ευχαριστω Ευχαριστώ και τον Ματιό Γκρός και τον Πατ Κόξ. Ποιος θα μου το έλεγε αυτό Κάποιο. Όταν τη περασμένη θητεία συζητούσαμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και καταθέσαμε και τροπολογία όπου θέλαμε να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στους συντονιστές των διαδρόμων, που θα μου το έλεγε ότι θα ήταν ο Ματιέ Γκρός ο, επόμενος ή ένας από τους ε, συντονιστές. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες ε, όσους θα θέλαμε ε, και τι να κάνουμε, δεχτήκαμε τους περιορισμούς που έχετε εσείς στη δουλειά σας, άρα και τις δυσκολίες. Τούτων λεχθέντων, όταν συζητήσαμε για τα διευρωπαϊκά δεκτία, ορίσαμε τα έργα με πολύ συγκεκριμένους όρους. Πρώτον, θα πρέπει να είναι έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και επιγόντως θα πρέπει να ε, βλέπαμε, λέγαμε, τις παραμεθόριες περιοχές γιατί εκεί είχαμε προβλήματα. Και κυρίως επειδή μας κόστιζε ετησίως το 1% του ΑΕΠ μας στην Ευρώπη. Το να μην έχουμε ε, συντονισμό, να είναι τόσα τα φορτηγά που να πηγαίνουν έρχονται στα σύνορα. Ερώτηση λοιπόν πρώτη. Μιλούμε για την εκτέλεση των έργων και για την ανάλυση ε, κόστους ωφέλειας, ε, για την εκτέλεση και την υλοποίησή τους. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα κάνετε και ανάλυση ωφέλους για τη μη εκτέλεση των έργων αυτών ή για την εκτέλεση ορισμένων που είναι μισοτελειωμένα, που έχουν φάει ένα σκασμό λεφτά από ε, χρηματοδότηση, αλλά που δεν καταλήγουν πουθενά. Δεύτερον, θα πρέπει να διατηρήσουμε τη συνοχή σε όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε και όλες τις ευθύνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το διαγωνισμό. Τα κράτη-μέλη έχουν καταθέσει λίστες προγραμμάτων, έργων και αν δεν τηρήσουμε αυτά τα κριτήρια, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προτεραιότητα στη μεθόριο, θα υπάρξει πρόβλημα. Σας ερωτώ, τι δυνατότητα νομίζετε ότι έχετε να πιέσετε τα κράτη-μέλη και να τα επηρεάσετε στη στιγμή της επιλογής των έργων. Από τα έργα που κατέθεσαν δηλαδή και θα επιλεγούν κάποια για να τα εκτελέσουν σύμφωνα ε, με το χρηματοδοτικό μέσο. Εσείς έχετε καμιά δυνατότητα να πείτε ότι αυτό το έργο δεν είναι προτεραιότητα και θα πρέπει να δούμε τι θα εφαρμόσουμε σύμφωνα με τις λιμένες αποφάσεις. Και μια τελευταία παρατήρηση. Πρόσφατα διαβάσαμε ότι έχουμε το, το πιο γρήγορο, λέει, τρένο υψηλής ταχύτητας που μπορεί να φτάσει την ώρα 581 χιλιόμετρα. Όχι στην Ευρώπη, αλλά στην Ιαπωνία. Και μιλάμε και για τρένα ε, ε, μαγνητικής ε, ανύψωσης. Οσάκα, Τόκιο που είναι 500 χιλιόμετρα το κάνει σε μία ώρα. Εμείς ως Ευρωπαίοι είμαστε ανίκανοι ε, σε κάποια μέρη της Ευρώπης να αντιμετωπίσουμε τρένα υψηλής ταχύτητας για να λύσουμε ένα πρόβλημα διαμεθοριακό. Δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Και ποιους λίντερ, ούτε ηγέτες θα είμαστε ούτε πουθενά. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ομό, αλλά έτσι θα βλέπω τα πράγματα να κάνουμε μια παγκόσμια ανάλυση. 500 χιλιόμετρα την ώρα πάνε οι άνθρωποι με, με, τρένα που πετάνε, μαγνητικά, με διπλώματα εύρεση τεχνίας που κάνουν έρευνα παγκόσμια οι άνθρωποι εκεί. Διπλώματα εύρεση τεχνίας που για μας είναι επιστημονική φαντασία. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει και έλλειψη αποφασιστικότητας, ηγετησίας της Ευρώπης δεν ξέρω, κάπως θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Έχουμε αυτό το εργαλείο που ονομάζεται Shift to Rail, αλλά δεν φτάνει ούτε κατά διάνοια στους Ιάπωνες. Και ό,τι διαβάζω, θα πρέπει να αρχίσουμε να αγοράζουμε τις πατέντες, γιατί μας έρχεται πιο φτηνό από ότι να κάνουμε έρευνα στην Ευρώπη και να βγάλουμε δικές μας τεχνίες. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει στον κόσμο. Ευχαριστώ, Γιάννης Νίλσεν. Eh, Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε το όραμα, έχουμε τα εργαλεία, αλλά πρέπει να γίνει και η δουλειά. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε την απόφαση που πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη κλπ. κλπ. Αλλά μιλήσατε και για το ρόλο των περιφερειών και αυτό το είπαμε λίγο σύντομα. Ενώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι περιφέρειες πρέπει να κινητοποιηθεί και ο κάθε δήμος και κοινότητα και ολόκληρη η οικονομική ζωή εκεί να αλλάξει. Επίσης, οι περιφέρειες μπορούν να πιέσουν το κεντρικό κράτος και τις αρχές και γι' αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Παύλ Τερίτσκα. Uh, uh, uh, Καλό σας απόγευμα. Εφήγησαν πολλά ζητήματα που μας απασχολούν. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο ζητήματα, δύο ερωτήσεις. Ένα από τα ζητήματα που μου έκαναν εντύπωση είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, που οι Ευρωπαίοι συντονιστές είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές ε, μέσω διαδρόμων, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε την προστιθέμενη αξία ε, ορισμένων, μιας μορφής μάλλον ή μορφών μεταφορών έναντι άλλων. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα δηλαδή. Και κύριε Γκρός, είσαστε υπεύθυνο για ένα διάδρομο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είμαι Τσέχος και μίλησα και με τον Υπουργό Μεταφορών που αντίθετα με τους προκατόχους του ενδιαφέρεται και για τις πλωτές μεταφορές. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Εάν λάβουμε υπόψη το διάδρομο που σας απασχολεί εσάς που με ενδιαφέρει και μένα, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία στη, ως προς τη χρήση των πλωτών ε, μεταφορών σε σχέση με άλλους, άλλες μορφές μεταφορών, ιδιαίτερα στις ε, ορεινές περιοχές. Στον πρώην διάδρομο που είχε συμφωνηθεί, συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο, τον δέχτηκαν τα κράτη-μέλη, αλλά στην πράξη αρκεί ένα κράτος να μην συμφωνήσει ε, για να τεθούν σε ομοιρία όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε χρηματοδοτικά μέσα, όχι πάντα επαρκή. Μπορούμε για τα ε, μικρότερα κράτη-μέλη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν έχουν ε, απόλυτα προσδεθεί στο άρμα των μεταφορών. Ε, και σε αυτή την περίπτωση αρκεί ένα κράτος να μην κινείται αρκετά γρήγορα για να αποδυναμωθεί το όλο σχέδιο πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή Μεταφορών, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να δούμε και στο μέλλον. Μαρία Γκραπίνη, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, τους συντονιστές και τώρα που μας παρουσίασαν αυτό το πλαίσιο όλα είναι πιο διάφανα Ε, αυτό που με ενδιέφερε ήταν από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Αλλά μου ελέγχθη ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πηγή χρηματοδότησης ε, για τις συνδυασμένες μεταφορές πάντα. Μπορείτε να μου πείτε από πού θα προέλθουν τα χρήματα και πόσα θα είναι ακριβώς αυτά. με ανησύχησε αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος Γιούνκερ αρκετές φορές ως προς την επιλογή των ε, σχεδίων από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια των ε, προγραμμάτων επενδύσεων γιατί δεν μπορούν να συμπεριληφθούν και οι 11 διάδρομοι παράλληλα. Ποια είναι τα κριτήρια. Γιατί ε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς θα ελέγξουμε και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έξι ανθρώπους που ελέγχουν το όλο πλαίσιο χωρίς ε, να υπάρχει κανένας έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια συνδεσιμότητα των σχεδίων. Πώς θα διαχειριστούμε αυτά, αυτούς τους διαδρόμους, ιδιαίτερα όταν είναι διασταυρούμενοι οι διάδρομοι. Ας πούμε, ε, τι θα γίνει όταν ένα κράτος ε, βάζει διόδια ή τέλη που είναι πολύ υψηλότερα από μια άλλη χώρα, γειτονική χώρα για το ίδιο δίκτυο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θέλω να αναφέρω τα δύο εξής την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, το λέω πολύ συχνά, είπες ότι ε, το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη είναι κουρελού και μάλιστα τρίπια στα σύνορα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ερφούρτη Ρεμβέργη, 20 χρόνια κάνουμε τρένο στην ε, ε, Γερμανία με ένα δισεκατομμύρια, αλλά από το Μόναχο μέχρι τη σύραγγα του Μπρένερ ε, στα σύνορα δεν έχουμε λόγο, έχουν κλείσει και τη γραμμή και αυτά είναι μεγάλα έργα τελείως ε, ε, μεταξύ του ασύνδετα. Ο Ματιό Γκρός αναφέρθηκε και στις μικρές διασυνοριακές συνδέσεις. Βερολίνο-Βρότσλαβ έχουμε σταματήσει ένα τρένο τώρα γιατί λείπουν 100 εκατομμύρια. Ναι, 100 εκατομμύρια σημαίνει δύο ώρες λιγότερη ε, ε, διαδρομή. Γιατί θα συνέφερε να παίρνει το τρένο και ε, όχι το πούλμα, το λεωφορείο. Αυτά τα 100 εκατομμύρια δεν τα έχουμε στη Γερμανία. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Τγάρδι Ούλμ δίνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να κερδίσεις ένα τέταρτο ή 30 λεπτά. Με... 400 εκατομμύρια, 12% είναι η χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι ανόητες κινήσεις. 400 εκατομμύρια δίνουμε ε, για ένα τέταρτο και δεν βρίσκουμε τα 100 που θα μειώσουν τη διαδρομή κατά δύο ώρες. Το 90% των ε, επιβατών στο σιδηρόδρομο είναι για μικρές αποστάσεις κάτω των 50 χιλιόμετρων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα μεγάλα έργα. Και άμα είναι 30-40 χρόνια ε, τα συνεχίζουμε τα έργα και είναι εις βάρος των μικρών. Το δεύτερο ερώτημα, ανάλυση κόστους ωφέλειας. Εγώ που ασχολούμαι 30 χρόνια με τις μεταφορές έχω την εξής εμπειρία. Αυτό που θέλει η πολιτική το το κάνει να, είναι, να φαίνεται φθηνό και αυτό που δεν θέλει το κάνει να φαίνεται ακριβό. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Το εξή ένα. Πριν από 25 χρόνια ξεκίνησε ε, η υπόθεση της Στουτγάρδης 21 για τον, ε, για τον σιδηροδρομικό σταθμό. Έλεγαν ότι θα πουλήσουμε το οικόπεδο ε, για να κάνουν μαγαζιά και θα χρηματοδοτήσει τη βήθηση του σιδηροδρόμου που θα γίνει υπόγειος και τώρα έχουμε 7 δισεκατομμύρια κόστος. Γύρω από τη Δρέστη ε, ε, φτιάξανε ένα δακτύλιο κλειστό, χωρίς να μπαίνει ούτε να βγαίνει κανείς. Και βγήκε ένα κόστος ωφέλεια θετικό. Εγώ δεν χρειάζεται να είμαι μηχανικός, ούτε συγκοινωνιολόγος, ούτε να έχω λεφτά, ούτε να μην έχω για να το απορρίψω. Αλλά το προβάλλουν θετικά αυτοί. Και χτες διάβασα μία ανάλυση για το νέο του, τούνελ της στο Ζέμεριν. Ε, από το μόνο ένα γραφείο έκανε την ανάλυση που σύμφωνα με τα κριτήρια τους είπαν ότι αν ε, φτιαχτεί αυτή η Ιραγκά και ξανακλείσει αμέσως έχουμε θετική ε, έκβαση 1,4% ωφέλεια. Αυτό εντάξει θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά ε, δεν είναι καλό έργο. Αυτό που υπολογίζουν ε, και αυτό που είναι αποφασιστικό για εκείνους που σχεδιάζουν τα έργα είναι η ίδια η κατασκευαστική δραστηριότητα και πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται την ώρα που χτίζεται το έργο και ε, το, μετά δεν τους ενδιαφέρει. Και λείπουν και τα κίνητρα. Τα κράτη-μέλη τυφλώνονται μόλις φτάνουν στα σύνορα, δεν βλέπουν παραπέρα. Ε, και πού είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και εγώ δεν μιλάω για 40-50%. Μας λείπουν μικρά κομμάτια από ε, τα σύνορα μέχρι τον επόμενο συνδρομικό κόμβο. Εκεί να είναι η χρηματοδότηση και με τη συνοχή και με τα διαρθωτικά μέχρι το 85%. Δεν είναι πολλά λεφτά, γιατί είναι μικρά τα διαστήματα, 10 χιλιόμετρα ξέρω εγώ, 5, ε, 8. Αυτό θα είναι η πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και ποια δυνατότητα βλέπετε εσείς να αλλάξει. Ε, βγαίνει και λέει ο Γερμανός υπουργό Μεταφορών, δεν έχω λεφτά, μου δώσετε ευρωπαϊκά, θα το κάνω. Και θα είναι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, πριν όμως απαντήσετε, θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπω δεν θέλει να μιλήσει καθόλου. Δεν θέλει, δεν θέλει, μια χαρά. Ωραία, έχουμε και το χρόνο μας. Δεν ξέρω ποιος θα αρχίσει, συμφωνήστε, βρείτε τα. Ο Πατ Κόξ. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Θα αναφερθώ σε μερικές και θα δούμε, Ματιέ, πώς θα χειριστούμε τις υπόλοιπες. Μιλήσατε για το ΕΦΣΙ, πολλοί από εσά, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ας αρχίσω από αυτό. Όπως και εσείς περιμένουμε τις ε, λεπτομέρειες του κανονισμού που διέπει το Ταμείο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα προτείνουμε αναδιάδρομο ε, να εξετάσουμε όλα τα σχέδια, τα προγράμματα και να δούμε ποια είναι τα πλέον συνεπή, δηλαδή που συνάδουν με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση αυτού του επιπρόσθετου Ταμείου. Ε, βεβαίως ε, δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα, δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία, θα δούμε τις λεπτομέρειες του κανονισμού. Θέλουμε όμως να κάνουμε την καλύτερη χρήση του εύση τη στιγμή που υπάρχει. Από το διάλογό μας με την ΕΤΕ, πριν ακόμα... Με την ΕΚΤ, με συγχωρείτε, πριν ολοκληρωθεί ο κανονισμός, ε, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να αποσβέσουμε αυτά τα σχέδια και τα προγράμματα τη στιγμή που έχουν ένα κύκλο ζωής και θα πρέπει να επιστρεφούν, επιστραφούν οι δαπάνες. Δηλαδή μιλάμε για, ένα, για μια κοινωνική επένδυση κεφαλαίων αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ορισμένα σχέδια δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες που διέπουν το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν προτρέχω, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Η ΕΤΕ στο διάλογο με τους συντονιστές, στο διάλογο μας, είπε ότι θα προσπαθήσει να ορίσει ένα σύστημα προώθησης των ομολόγων έργου δηλαδή ε, θα λάβουμε υπόψη ε, λίγο υψηλότερους ε, κινδύνους από αυτούς που είναι οι μέση κίνδυνοι και αυτά τα σχέδια θα χρηματοδοτηθούν εν μέρη. Και έτσι θα είχαμε μία ομολογία έργου σε χαμηλότερο κόστος και με καλύτερο rating με καλύτερη αξιολόγηση. Έτσι θα λειτουργήσει έμπρακτα. Πολύ μιλήσατε για τη, τα ομόλογα έργου, τα πιλωτικά ομόλογα έργου. Ε, τα χρόνια αυτά που συντονίζω αυτές τις εργασίες μπορώ να σας πω ότι καμία τέτοια ομολογία έργου δεν έφτασε μπροστά μου. Άρα καμία ομολογία έργου δεν αφορά ε, ένα πρόγραμμα μεταφορών το οποίο με απασχόλησε μεν. Ο κύριος Ρικέ μίλησε για 30 δις και είπε ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτω από 10. Μπορώ να σας πω ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά 12 δις. Και όπως είπε και ένας συνάδελφός σας, αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ε, αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου υψηλού ενδιαφέροντος στις τάξεις του 3 1. Και ως προς τους οριζόντιους διαδρόμους υπάρχει ενδιαφέρον της τάξης 10 προς 1. Ρωτήσατε ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα κάνει την αξιολόγηση για να δούμε το ε, CEF. Υπήρχε εξωτερική αποτίμηση όπου ε, έγινε μια συγκεκριμένη στάθμιση για να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τον κανονισμό, σε σχέση με τους συνδέοντας στην Ευρώπη. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι καθεστώς αδειοδότησης θα υπάρξει. Ξέρω ότι έχει προχωρήσει αυτή η εργασία. Μετά θα έρθει στην ΙΝΕΑ, δηλαδή στον οργανισμό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρατηρήσεις και σε κάποια φάση οι συντονιστές στη συνέχεια θα δουν πώς ναι. έχουμε προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περιμένουμε, κρατάμε στάση αναμονής δεν θα γίνει η απότερη κρίση με βάση ένα συγκεκριμένο κανονισμό, αλλά οπωσδήποτε θα λάβουμε υπόψη μαζί σας τις δυνατότητες που μας δίνουν οι κανόνες. Τώρα, σε σχέση με τα ε, κεντρικά δίκτυα ή διάφορες υποδιαιρέσεις τους, δεν το αποφασίσαμε εμείς. Όπως και εσείς ε, ψηφίσατε για ένα παρά παράρτημα και το οποίο μας δώσατε πίσω. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που αποφασίζουν, που καθορίζουν την γενικότερη πολιτική. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό δόγμα από τις ε, Βρυξέλλες. Υπάρχει ένας διάλογος και έτσι προωθούνται τα ζητήματα. Τώρα για να επανέλθω στο θέμα της χρηματοδότησης, ένα από τα ζητήματα που θίξατε πολλοί από εσά, αφορά τα 2,7 δις που θα φύγουν από το συνδέοντα στην Ευρώπη ε, μέσα στα πλαίσια της κεντρικής χρηματοδότησης του σχεδίου ε, Juncker. Το CF, το συνδέοντα στην Ευρώπη, αφορά μια γενικότερη αποτίμηση που θα γίνει το 2016. Επειδή λοιπόν γίνεται ε, μπροστομερής χρηματοδότηση, θα μπορέσουμε να έχουμε μία αντιστοιχία τελικά και στη δεύτερη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπήρχε πολύ, μικρότερη, πολύ μικρότερο ποσό από το αν δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο πρώτο σχέδιο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 2,7 δις που εντάσσονται στο σχέδιο Juncker από τα 12 ε, δις. Δεν ξέρουμε όμως αν θα χάσουμε ε, χρήματα από την πίσω πόρτα με το σχέδιο Juncker και τα πάρουμε από την προστινή πόρτα χρησιμοποιώντας το σχέδιο Juncker. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι οι υποδομές μεταφορών στις περιφέρειες για να έχουμε μία κατάσταση συνολικού κέρδους, διότι δεν ξέρουμε ε, ποια θα, ποιες θα είναι τελικά οι πηγές εσόδων με βάση τις ομολογίες έργου. Μιλήσατε για τη σχέση κόστους-οφελίας. Ποια επιτόκια θα χρησιμοποιήσουμε όταν έχουμε ε, μειώσει εκπτώσεις έτσι ώστε να έχουμε μία συνολική απόσβεση. Αυτό θα το δούμε κατά περίπτωση και θα δούμε πώς ε, οι εθνικές κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Δεν θέλω να μιλήσω για το δικό μου διάδρομο τώρα, αλλά πολλά θέματα του δικού μου διαδρόμου που αφορούν τη Γερμανία περιμένουν τις ε, αποφάσεις από το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών μέσα στα πλαίσια της προτεραιότητας επενδύσεων. Άρα, ως προς το δικό μου διάδρομο, μπορώ να πω ότι πολλά ζητήματα δεν τα ξέρω γιατί περιμένω τις αποφάσεις των ε, γερμανικών αρχών. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε μία γενικότερη όθηση σε αυτά τα σχέδια με βάση ένα συγκεκριμένο χρονισμό ως προς το ERTMS και θα σταματήσω εδώ το θέμα που, ε, στο οποίο αναφερθήκατε αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης τη Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας. Ο κύριο Βίνκ είπε ότι προσπαθεί ο συντονιστή να δει χιλιομετρικά πώς μπορεί να λάβει υπόψη μικρότερε μικρότερες αποστάσεις που αν μεταφερθούν σε όρους ERTMS θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη συνδεσιμότητα. Δηλαδή να έχουμε μικρότερα ε, κομμάτια του συστήματος που θα δώσουν ε, μια καλύτερη διαλειτουργικότητα διασυνοριακά. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, γίνονται και αν γίνονται διακρίσεις ως προς την ανταπόκριση των κρατών ε, μελών. Αν υπάρχουν διαφορές. Για το δικό μου ε, διάδρομο έχω 7 κράτη-μέλη συν την Νορβηγία. Και όλες οι χώρες έχουν εγκρίνει τα προγράμματα. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα προγράμματα. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν υπάρχουν ε, σοβαρές διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών ή συντονιστών σε σχέση με, τη, με τις γενικότερες ιδέες που διέπουν το σχέδιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μία επενδυτική ευαισθητοποίηση από πλευράς οι e Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο-τρία χρηματοδοτικά συγκεκριμένα. Για το χρόνο πόσβεσης, Ξέρουμε βεβαίως ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, δεν το παραγνωρίζουμε. 25 χρόνια σε σχέση με κάποιες υποδομές είναι όντως παράλογο διάστημα και η μελέτη που αναφέρθηκε ακριβώς αυτό εξετάζει. Αν δούμε πότε αρχίζει να αποδίδει μία επένδυση, θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες οι προθεσμίες και οι διάρκειες από ό,τι ε, ακούμε. Το δεύτερο αφορά την ανάλυση του Ντομινίκ Ρικέ. Έχει απολύτως δίκιο, 100%. Σε ό,τι αφορά τα έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, όποιος χρησιμοποιεί σήμερα αυτό το ταμείο δεν προσανατολίζεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της δικές μας των δικτύων. Βλέπε σιδηρόδρομο, βλέπε εσωτερική ναυσιπλοεία κτλ. Άρα στις μεταφορές ε, θα έχουμε ε, μετατόπιση του κέντρου βάρους ή μετατόπιση της χρηματοδότησης. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο. Για μένα η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη είναι προστιθέμενη αξία για το λεγόμενο σχέδιο Juncker, αλλά δεν πρέπει αυτά να ειδωθούν ούτε ανταγωνιστικά ούτε ως υποκατάστατο. Μόνο από κοινού για να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα από όσα ελπίζουμε αυτόν τον καιρό. Τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ το μέλλον του Ταμείου Στρατογικών Επιδίσεων. Τα ομόλογα έργου αξίζουν τον κόπο και τα είπε και ο κύριος Ρικέ και τα γνωρίζει πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει βγάλει μια έκθεση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τα τρέχοντα έργα, είναι 7 τον αριθμό, ε, με ομόλογα έργου και διαπιστώνεται ότι ε, τα έργα που αξιοποίησαν αυτά τα ομόλογα έχουν μια μοχλευσή της τάξης του 1 ε, επί 30 αν είναι καλά τα έργα και προσφέρονται, είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα ομόλογα έργου και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αλλά επαναλαμβάνω, το ΕΦΣΥ δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει το σιδηρόδρομο ανάμεσα σε δύο χώρες, ούτε πρόκειται να επισκευάσει το δίκτυο. Ε, Έχουμε ένα διάδρομο που συγκεντρώνει εννέα χώρες, το δικό μου, ε, και είναι πολύ καλή συνεργασία, αλλά η ώρα της αλήθειας δεν είναι ακόμα τώρα. Είναι όταν θα αρχίσει η υλοποίηση των έργων. Γνωρίζω ότι όχι μόνο στο δικό μου διάδρομο και σε άλλους η σύνδεση μεταξύ δύο κρατών είναι και παραμένει αγκάθη. Αλλά ως συντονιστής και να δανειστώ μία ρίση του κόξ, εμείς είμαστε συντονιστές, δεν είμαστε ε, δικτάτορες. Δεν θα επιβάλλουμε στη χώρα τι θα κάνει, συντονίζουμε. Λέμε ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ, δεν πρόκειται με το ζόρι να του επιβάλλουμε τι έργο θα κατασκευάσουν. Είχα πάει εγώ στα σύνορα Γερμανίας Τσεχικής Δημοκρατία, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί κανεί να πιέσει και να πει είναι πολύ σημαντικό να μην έχετε μόνο ε, τα εθνικά γυαλιά αλλά και τα ευρωπαϊκά, να βλέπετε την κατάσταση ευρύτερα. Ε, και αποδίδουν και αυτά τα λέμε. Υπάρχουν και οι δυνατότητες και τα μέσα για να πιέσουμε και για να αποδείξουμε ότι αξίζουν τον κόπο κάποιες επενδύσεις. Αν όχι βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον μέσο πρόθεσμα. Από πλευράς μεθόδου λοιπόν και τα κράτη έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Αλλά είναι πολύ θετικές οι ειδήσει αν δω μια χώρα όπως η Γερμανία, Γκεζινέα, από που περνάνε έξι διάδρομοι, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν ήταν μόνο ε, η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και σημαντική εταίροι όπως είναι η γερμανική σιδηρόδρομη, όπου έχουν ε, συζητήσει με τους συντονιστές έξι διαδρόμων. Και αυτό το παράδειγμα ε, δημιούργησε σχολεία, που πούμε, και το μιμήθηκε και η Γαλλία, υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών και στο εσωτερικό των κρατών, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις. Τι θα ακολουθήσει τώρα αυτό θα είναι η ώρα της αλήθειας. Για την οικονομία και την οικολογία και πώς θα το συνδυάσουμε. Τα ξέρετε αυτά. Πώς εργαζόμαστε, ρώτησε η κυρία Καρυμαντελή, πολύ συγκεκριμένα. Πήγα και στη Δρέσδη και στην Πράγα και είπα ότι θέλω να δω όχι μόνο τους υπουργούς, από τους που με δέχτηκαν, εντάξει, όχι μόνο τους ε, ε, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς, αλλά και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ. του είδα και τους ρώτησα, εσείς θέλετε να συνεργαστείτε, ε, είστε εδώ για να μας βοηθήσετε να κάνουμε τη γέφυρα μεταξύ οικολογίας και οικονομίας ή απλώς να καταγγέλλετε και εξεπλάγει θετικά γιατί ήταν θετική η ανταπόκριση. Δεν θέλω να το κάνουν μόνο στη χώρα τους, αλλά να βοηθήσουν και σε μια υποδομή, σε μια δομή που θα έχει ε, διασυνοριακή μορφή φερρυπίν. Ε, αυτά μπορούμε εμείς να τα κάνουμε, αλλά και σε εμά εναπόκειται να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Τι γίνεται με την εσωτερική πλοία, Σε ορισμένες περιφέρειες πρέπει να κάνουμε επιλογές. Και απαντώ στην ερώτηση του Βιμ Βαντενκάμπ, ε, ε, είμαι υπέρ ε, της συνοριακή και διαλειτουργικότητας, αλλά σήμερα οι μεταφορές είναι κατά 80% οδικές. Εάν δεν βρούμε εναλλακτική λύση, αυτό θα είναι εις βάρος πολλών περιφερειών και πολλών επενδύσεων. Εμείς γνωριζόμαστε καλά από το παρελθόν. Εγώ δεν είμαι δογματικός, ε, ούτε άκαμπτος. Θα το επιλέξει η οικονομία. Ας μην γελιόμαστε βήμα, ότι συμφέρει περισσότερο τον κλάδο. Ε, αλλά μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε τις υποδομές και αυτό θα βελτιώσει τη ζωή και των ανθρώπων επιτόπου και την οικονομία. Αυτή η διαλειτουργικότητα, οι συνδυασμένε μεταφορές είναι κάτι που το έχουμε αρχή μας, αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε θα το, όταν δεν το θέλει ο κόσμος, όταν δεν το θέλει η πολιτική. για τον ποταμό Έλβα, ας πούμε, λέμε ότι εδώ, ορίστε, έχουμε μεταφορές ανάμεσα σε δύο πόλεις. Ε, ε, ε δεν γίνεται ε, αυτό με το σιδηρόδρομο, δεν γίνεται με τον αυτοκινητόδρομο. Ε, τι θα γίνει λοιπόν, θα παραμείνει αυτός ο κλάδος, ε, δημιουργεί και θέσεις εργασίας, θέλουμε να παραμείνει, γιατί χρειάζεται αυτές οι μεταφορές. Αλλιώς θα πούμε ότι αυτός ο κλάδος έχει πεθάνει και ωραία, να δούμε κάτι άλλο. Τι γίνεται όμως με τις θέσεις εργασίας και τους ανθρώπους που εργάζονται. Αυτό είναι το θετικό ως προσέγγιση. Όταν λες ότι θέλω ή δεν θέλω ένα μέσο μεταφοράς για διάφορους λόγους, αυτό συνδέεται με ανθρώπους, με περιφέρεια, με ανάπτυξη, ε, με την κινητικότητα ολόκληρη της περιοχής. Τελευταία. Νομίζω απάντησα για τον Έλβα και την αποτάμια Για την ψηφιοποίηση. Βεβαίως, για μας η ψηφιοποίηση είναι και παραμένει ένα θέμα και μια πρωτοβουλία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσο και σημαντική. Και το να δημιουργείς ε, διευρωπαϊκά δίκτυα δεν σημαίνει ότι χτίζεις καινούριες υποδομές παντού. Ε, σημαίνει και βελτιστοποίηση, βελτίωση, επισκευή υφισταμένων δικτύων και υποδομών. Υπάρχουν υποδομές. Πρέπει να καταργήσουμε και άλλα εμπόδια. Εάν επενδύσουμε σε μια περιφέρεια για να μειωθεί κατά δύο ώρες ε, μια διαδρομή. Τι να το κάνω αυτό μέσα σε μια χώρα αν φτάσει στα σύνορα και μετά πρέπει να περιμένει 7 ώρες για λόγους διοικητικού και τελωνιακούς. Ε, και εκεί μπαίνει η ψηφιοποίηση. Και σε πολλά προγράμματα, σε πολλά έργα δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. εγώ ξέρω στην Ευρώπη περιπτώσεις και λιμάνια ε, που η ίδια ε, δομή, η ίδια υποδομή με την ψηφιοποίηση μπορεί να διπλασιάσει τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα που μπορεί να δεχτεί. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι και διοικητικά και οργανωτικά. Δεν είναι μόνο τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το είπαμε στο παρελθόν. Για το σιδηρόδρομο Ακόμα στην Ευρώπη ο σιδηρόδρομος δεν είναι καθόλου ευρωπαϊκός, είναι ένα άθροισμα ε, εθνικών σιδηροδρόμων και εύχομαι καλή τύχη στο τέταρτο πακέτο ε, των σιδηροδρόμων και χωρίς να είμαι απεσιόδοξος μπορώ να προβλέψω ότι θα υπάρξει και πέμπτο και έκτο. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει ο Ευρωπαϊκός Σιδηρόδρομος και αν δεν ασχίσουμε ε, πίεση τότε χωρίς να, αυτό να είναι ένα κακό λογοπαίγνιο θα χάσουμε το τρένο αφού το έχουν καταφέρει άλλες τομές ε, ε, ε, στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε στην Ιαπωνία. Πριν από λίγους μήνες είχαμε κάνει εδώ μια εκδήλωση και ήταν και ο πρόεδρος των Ιαπωνικών σιδηροδρόμων και έλεγε ότι οι καθυστερήσει κατά μέσο όρο είναι 0,20 δευτερόλεπτα. Ναι, και σε μας έτσι είναι. Εμάς ούτε, ούτε το μετράμε. Κάτω από λιγότερα λεπτά δεν νοείται καθυστέρηση αυτό. Αυτά. Και ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο συγητές και συντονιστές μας που μας κάνατε αυτή την παρουσίαση και με χαρά περιμένουμε και τις επόμενες εκθέσεις όλων των συντονιστών ε, και των 11. Θα τα ξαναπούμε τότε. Ευχαριστώ πολύ και χαίρετε. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Also, klar. Πάμε στο επόμενο θέμα, στη διαταξή. Παρακαλώ τα πηγαδάκια εκτός της αιθούσης. Also, wir kommen Λοιπόν, επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπρένερ, εκτελεστικό διευθυντή του Eurocontrol. Θα μας δώσει μια ε, συνέχεια της συνέντησης που είχαμε στις 3 Σεπτεμβρίου. Ε, είχαμε συζητήσει, είμαστε για την Ουκρανία και για το πώς ε, απειλείται από στρατιωτικά αεροσκάφη πολιτική αεροπορία και άλλα θέματα συνεργασίας που μας απασχολούν και που έχουν να κάνουν με το μελλοντικό ρόλο της Eurocontrol του ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Κύριε Μπρένερ, έχετε το λόγο για 15 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ για τα ευγενικά σας λόγια. Εξέχοντα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά η ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για το τι συνέβη από την προηγούμενη φορά που είχα έρθει για να βελτιωθεί η ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές συγκοινωνίες. Ιδίως για τις πτήσεις πάνω από τη θάλασσα. Το Eurocontrol είναι μια διακυβερνητική οργάνωση 41 κρατών από την Ιρλανδία μέχρι την Αρμενία ή από την Πορτογαλία μέχρι την Εστονία. Εσθονία. Η Ουκρανία επίσης είναι μέλος του Eurocontrol. Uh, an EU body. Δεν είναι ενωσιακό όργανο, αλλά έχουμε μια συμφωνία υψηλού επίπεδου με την Ένωση από το 2013 και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά όργανα όπως την ΙΑΖΑ ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία με τα οποία έχουμε κοινά προγράμματα. Είμαστε πολιτικοστρατιωτική οργάνωση που συντονίζει στενά τις ανάγκες της πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας. Μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Network Manager και ο εδώ Network Manager λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για να ελέγχει την κυκλοφορία, ενέργεια κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται γιατί συνεχώς αυξάνονται οι αριθμοί των πτήσεων. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου των πτήσεων λοιπόν είναι κάτι στο οποίο θα επανέλθω μετά. Εδώ βλέπετε τους αεροπορικούς διαδρόμους. Όσο πιο παχύ το χρώμα, όσο τόσο πυκνότερη και η τόσο μεγαλύτερη αριθμή πτήσεων. Στην Ουκρανία και ανατολικά της σημειώθηκαν μερικές σημαντικές αλλαγές. Βλέπετε εδώ τις δύο γραφικές παραστάσεις διπλα Η διαφορά είναι ότι από τα γεγονότα της Κρυμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας υπάρχει συμφόρηση και απομακρύνεται η κυκλοφορία από την Ουκρανία μετατίθεται στην Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μειώνεται η κυκλοφορία στην Ουκρανία και στην Μολδαβία που δεν συμμετέχει ακριβώς σε αυτή την πυκνότητα αυτό έχει οικονομικές επιπτώσεις για τις χώρες αυτές. Και αρνητικές και θετικές, ή μάλλον ή αρνητικές ή θετικές. Γιατί η περισσότερη κίνηση σημαίνει περισσότερα κέρδη. Και άρα και περισσότερη δραστηριότητα των ε, ελεγκτών εναερίου κυκλοφορίας. Εδώ βλέπετε τους αριθμούς για το 13 και 14 τις παραστάσεις. Ανάλογες αλλαγές έγιναν και όταν άνοιξε το κοτσιφοπέδιο μετά από τα 15 έτη κλεισίματος του Αεριου χώρου του λόγω των πολέμων στα Βαλκάνια. Τώρα έχει ξαναρχίσει η εναέρια κυκλοφορία και πάνω στο κοσυφοπέδιο. Αυτό κάνει λοιπόν ο εναέριος ελεγκτής. Διαχειρίζεται τις πτήσεις και σε καιρό ειρήνης και σε καιρό σειράξεων ή διακοπής των πτήσεων. Γιατί σε αυτή την περίπτωση σειράξεων πρέπει οι πτήσεις να πετάξουν με διαφορετικό δρομολόγιο για να αποφύγουν το Γνωρίζουμε και την τελευταία καταστροφή και το κλείσιμο του εναερίου χώρου ολόκληρη τη Ανατολική Ουκρανία. Ο λόγο για τον οποίο κλείνει ένα εναέριο χώρο ε, αφορά τα κυρίαρχα έθνη και κράτη και η Ουκρανία αποφάσισε ότι θα ανοίξει ο εναέριος χώρος της αλλά μετά, στη, μετά από το τελευταίο γεγονός κλείσε θα σας πω όμως τι μπορεί να βελτιώσαμε. Οι χώρες γενικά χρησιμοποιούν μηνύματα που έχουν αυτήν τη μορφή. Εκδίδουν τις λεγόμενες νόταμς ή νότισης του έρμεν που δίνονται σε όλους τους χρήστες του εναερίου χώρου και δείχνουν ποιος χώρος είναι διαθέσιμος, ποιοι διάδρομοι και σε ποια ύψη και αν ο χώρος είναι ανοιχτός ή κλειστός. Αυτά διατίθενται 24 ώρες το 24 σε όλους τους χρήστες του χώρου. Και υπάρχει ένα, μια κεντρική τράπεζα δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και διατίθεται σε όλα τα χώρες μέλη της. Μετά το EAD λέγεται European Aeronautical Information System Database. Αλλά βέβαια τα διαδίδει μόνο με την άδεια των χωρών που ενδιαφέρονται. Οι χώρες λοιπόν μπορούν να εκδώσουν οδηγίες και εντολές ανάλογα με το αν είναι ανοιχτός ή κλειστός ο χώρος τους, μπορούν να το πληροφορούν αυτό στους χρήστες και μπορούν να δίνουν πληροφορίες στους χρήστες και άλλων χώρων αν πρέπει να τους αποφύγουν κλπ. Οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να απαγορεύσουν ορισμένες εταιρείες από την υπέρπτυση του χώρου της Ένωσης ή αν μερικών χωρών. Δεύτερον, οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν και αυτές μια ευθύνη λήψης αποφάσεων κάθε αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να αποφύγει κάποιον αεροπορικό χώρο ακόμη και αν θεωρείται επισήμως ανοιχτός από τη χώρα του. Χρησιμοποιεί διάφορα κριτήρια για τους διαδρόμους όπως το βάρος του καυσίμου, το κόστος των δασμών, τον καιρό και τελικά ως κριτήριο σε τι, ώρα θα φτάσουν στον προορισμό τους και φυσικά και το θέμα της ασφαλείας. Το μέγα θέμα λοιπόν είναι πώς μια χώρα ή κάποια εταιρεία μπορεί να πάρει την απόφαση αυτή, πώς αξιολογεί δηλαδή τον κίνδυνο υπέρπτυσης κάποιου χώρου. Και τώρα θα σας πω τι έγινε τελευταία. Όλοι καταλάβαμε ότι After group was. Με την πτήση MH17. Τι πήγε στραβά. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή μια αεροπορική εταιρεία ή ένα κράτος για την πτήση πάνω από χώρους σειράξεων. Τι πληροφορίες τις διατίθενται. Κάθε κράτος πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου ή κινδύνου ασφαλείας όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει στην επικράτειά της για να καταλήξει αν είναι ασφαλές ή μη ασφαλές να γίνουν πτήσεις στον αέριο χώρο της. Αυτό που δεν κάνουν όμως οι χώρες και που το εξετάζει η ΚΑΟ είναι αν, ότι δεν μοιράζουν τον χώρο. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι και άλλες χώρες θα έχουν αυτές τις πληροφορίες και όχι μόνο η σχετική νότα μου που σας ανέφερα πριν. Εδώ στο Safety Risk Assessment μιλάμε για τα βασικά στοιχεία που οδηγούν στην έκδοση μιας νότα μου. Καλό θα ήταν σκεφτήκαμε οι χώρες μέλη να του ζητήσουμε να συμμεριστούν τις αξιολογήσεις που κάνουν και για το γειτονικού χώρους και αυτό έγινε σε διάσκεψη της ΙΚΑΟ τον περασμένο Φεβρουάριο. Τα συμπεράσματα υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο της ΙΚΑΟ που απεφάνθη ότι σωστή είναι αυτή η πρόταση και έκανε επίσημη σύσταση τα κράτη να συμμερίζονται τις αξιολογήσεις τους. Αλλά δυστυχώς τα κράτη δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πληροφορίες για τον χώρο τους σε άλλες χώρες. Από την άλλη μεριά ήδη υπήρξε πίεση ώστε να χορηγηθούν τα στοιχεία και οι χρήστες του εναερίου χώρου θα βοηθούνταν ιδιαίτερα. Δεν είναι όμως οι χρήστες μόνο, είναι και γενικά οι άλλες χώρες που θέλουν να κάνουν αποτίμηση του κινδύνου για τις υπόλοιπες. Για να δουν αν θέλουν να έχουν το ίδιο συμπέρασμα με την χώρα που εξέδωσε το συμπέρασμα ή αν θα βγάλουν τα δικά τους. Έχουν γίνει πολλές φορές συζητήσει με βάση τη δημοσίευση στοιχείων αξιολόγησης του κινδύνου μεταξύ χωρών μελών, αν έχουν τα ίδια συμπεράσματα ή όχι. Καλό παράδειγμα ήταν πέρυσι, όταν τέθηκε το πρόβλημα της υπέπτυσης του αεροδρομίου του Τελαβίβ και οι Ηνωμένε Πολιτείες σταμάτησαν αμέσως τις πτήσεις τους προς το Τελαβίβ. Το Ισραήλ τότε πήρε την απόφαση να συμμεριστεί την ε, αξιολόγησή του και με βάση αυτή την αξιολόγηση και τις πληροφορίες που έδωσε η Άσα και η ΕΦΑΟ είπαν, ζήτησαν να γίνει υποχρεωτική η χορήγηση αυτών των safety risk assessment. Το Eurocontrol λοιπόν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται τις πληροφορίες τους αυτές, όχι μόνο με άλλες χώρες, αλλά και με το Eurocontrol που διαχειρίζεται το δίκτυο. 24 ώρες το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο. Όπως ζητάει η ΚΑΟ εξάλλου. Το Eurocontrol λοιπόν είναι ο διαχειριστής του δικτύου για τις 47 χώρες μέλη και έχει και δημόσιες και προστατευμένες μεθόδους για την χορήγηση αυτών των πληροφοριών. Στο προστατευόμενο δίκτυό μας δημιουργήσαμε ένα χώρο για την διαχείριση των κρίσεων και εκεί υπάρχουν νόταμ που αφορούν κλεισίματα αεναερίου χώρου από χώρες που απαγορεύουν ή συστήνουν στις αεροπορικές εταιρείε να αποφύγουν την υπέρπτυσή τους. Εδώ βλέπετε τι είδους κίνδυνοι υπάρχουν γύρω από την Ευρώπη. Η κατάσταση βέβαια δεν είναι στατική, ενημερώνεται συνεχώς και αλλάζει συνεχώς. Όπως σας είπα αυτά ενημερώνονται 24 ώρες το 24ωρο και τα δίνουν και όλοι σε όλους τους χρήστες του εναερίου χώρου. Άρα είμαστε όντως ένα κομβικό σημείο στη διαχείριση των εναερίων χώρων. Η ΙΚΑΟ έχει πάρει ορισμένα πρώτα βήματα να δημιουργήσει μια τράπεζα δεδομένων παγκοσμίως Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε συμπληρωθεί τελείως, αλλά μπορούν ήδη τα κράτη-μέλη να υποβάλουν πληροφορίες εκεί, ώστε να υπάρχουν τα στοιχεία και να διατίθενται. Αυτό βέβαια εθελοντικά για κάθε χώρα μέλος και η, η ΚΑΟ το συστήνει για ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η Ευρώπη βέβαια μόνο για τον εαυτό της. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ως Ευρωπαίοι την ΚΑΟ να πετύχει σε αυτήν τη σύστασή της. Επίσης, στον ιστοκόμπο μας προσθέτουμε και πληροφορίες που χορηγούνται από χώρες όχι μόνο για τον ίδιο τους τον χώρο αλλά και για χώρους άλλων χωρών μελών. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Μπορεί ένα κράτος να μην θέλει να χορηγήσει πληροφορία. Ή υπάρχουν κράτη που αποτελούνται από δύο διαφορετικές οντότητες ε, αντίπαλες και η νενομισμένη οντότης μπορεί να αντιτίθεται στη χορήγηση αυτών των πληροφοριών. Ή μπορεί δύο να είναι οι αναγνωρισμένες οντότητες και να δημοσιεύουν διαφορετικά στοιχεία. Με αυτή τη βάση φυσικά πρέπει να δούμε και τρίτες πηγές και όχι μόνο τι λέει μια χώρα και δημοσιεύει. Αυτό φυσικά είναι πιο ενδιαφέρον σε περιπτώσεις και σημαντικό σε περιπτώσεις σειράξεων. Οι πληροφορία μιας χώρας για την κατάσταση του χώρου μιας άλλης χώρας είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι ανάγκη να αποκαλύπτεται η πηγή. Πρέπει όμως να είναι χώρα η πηγή. Αυτό έχει βοηθήσει πολλές φορές για να αρχίσει ας πούμε συζήτηση ως προς το τι θεωρεί μια χώρα για την κατάσταση ασφαλείας μιας άλλης. Και αυτό που έχει σημασία είναι να προχωρήσουμε με βάση τις ε, πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ε, τη δημοσίευση ε, ενός δελτίου για το αν ε, μία διέλευση είναι ασφαλής ή όχι, αλλά και μία γενικότερη αποτίμηση των κινδύνων. Πιστεύουμε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εταιρεία που χρησιμοποιούν έχει πληροφορίες και ε, οι πληροφορίες αυτές ε, δεν θα αφορούν μόνο την ε, επωνομαζόμενη flag area. Θεωρούμε ότι όποια αεροπορική εταιρεία και να χρησιμοποιούν οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εταιρεία αυτή έχει τις ίδιες πληροφορίες, διαθέτει τις ίδιες πληροφορίες. Γι' αυτό ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας ε, ε, υποστηρίξει στην συμπλήρωση αυτών των ε, πληροφοριών και διάθεσή του στο δίκτυο μέσα στα πλαίσια μίας πλατφόρμας διανομής πληροφοριών ή δημοσιοποίησης πληροφοριών και στα 41 κράτη και να μπορέσουμε να είμαστε ένα ε, σημείο αναφοράς στην ε, συνολική ε, τράπεζα δεδομένων του ΙΚΑΟ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει τα κράτη να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με τον διαχειριστή δικτύου και να βοηθήσουμε την ΙΚΑΟ να έχει μια πολύ καλή τράπεζα δεδομένων, η οποία να στεφτεί από επιτυχία τώρα από το σενάριο κρίσης και την αποτίμηση κινδύνων μιλώ, θα μιλήσω για την εποπτεία ε, στις ανοιχτές θάλασσες. Τους τελευταίους μήνες ε, είδαμε ότι ε, έγινε μία εντατικοποίηση της εποπτείας στις ανοιχτές ε, θάλασσες. Η Ρωσία δεν είναι ένα από τα 41 κράτη της, του Eurocontrol και μετά την κρίση της ε, Κρυμαίας εμείς το Eurocontrol έχουμε παγώσει κάθε επαφή με τη Ρωσία. Πριν από την κρίση της ε, Κρυμαίας και την κρίση στην Ανατολική Ουκρανία. Είχαμε μια περιφερειακή συνεργασία με τη Ρωσία, όμως μετά από αίτημα ευρωπαϊκών κρατών θεωρήσαμε ότι το Μάρτιο έπρεπε να συγκληθεί σύσκεψη όλων των κρατών του Eurocontrol και της Ρωσίας για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στις ανοιχτές θάλασσες. Θεωρήσαμε λοιπόν Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε την ε, κατάσταση, να αποτιμήσουμε την κατάσταση σε σχέση με τις στρατιωτικές δραστηριότητες της ε, Ρωσίας και θεωρήσαμε ότι ε, οι προδιαγραφές του ΙΚΑΟ απορρέουν από το πρόγραμμα του 1960 όπου δεν υπήρχαν τόσο έντονες, ε, τόσο υψηλές ε, προδιαγραφές και τέτοια χρήση στις, ε, των εναέριων διαδρόμων στη, πάνω από τις ανοιχτές θάλασσες. Αυτό το εργαστήριο έφτασε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη βελτίωση της ΙΚΑΟ και το δεύτερο εργαστήριο ε, οργανώθηκε ε, φέτος τον Απρίλιο με την ΙΚΑΟ στο Παρίσι. Επιτελέστηκε πρόοδος και φτάσαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια αν έχουμε το πρόγραμμα, τα flight plans, τα το σχέδιο πτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τα σχέδια πτήσης και για τις ε, εμπορικές καθαρά πτήσεις, όχι δηλαδή τις στρατιωτικές. Ναι, και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει πλήρης αναγνώριση της πτήσης και κατά πόσο υπάρχει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο πτήσης. Η Ρωσία υποστήριξε αυτό το σχέδιο και είπε ότι μπορεί να υποβάλει τέτοια σχέδια πτήσης και γι' αυτό τώρα εργαζόμαστε σε τεχνικό επίπεδο για να λάβουμε αυτά τα σχέδια και για να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστή δημοσιοποίηση των σχεδίων πτήσης. Και αυτό αφορά όλα τα κέντρα εναέριας κυκλοφορίας. Βλέπουμε το, το χρόνο, το που βρίσκεται το αεροσκάφος και το ποια είναι η πορεία του. Στο παρελθόν είχαμε την ταυτοποίηση με βάση ε, συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία όμως δεν ήταν τόσο τελειοποιημένα. Εφόσον λοιπόν η Ρωσία δέχτηκε να ε, δημοσιοποιεί τα σχέδια πτήσης για τις εμπορικές πτήσεις, φτάσαμε σε συμπεράσματα στο εργαστήριο με την ΙΚΑΟ και μπορέσαμε να επικαιροποιήσουμε το πλαίσιο δράσης της ΙΚΑΟ έτσι ώστε και στο μέλλον να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα, ως προς τα ατυχήματα και τα συμβάντα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποτρέψουμε. Εάν όμως ε, επισυμβούν, δεν μπορούμε παρά να δράσουμε τάχιστα, αλλιώς θα ήμασταν ανεύθυνοι, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια των επιβατών για το μέλλον. Γι' αυτό χρειάζεται και στρατιωτικό συντονισμό. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει και η αποτίμηση κινδύνων σε ε, επίπεδο διαχείρισης διεθνών ε, κρίσεων ή στην εποπτεία πάνω από, τις, ε, από την ανοιχτή θάλασσα. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα της ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριε Μπρένερ. Τώρα έχουμε πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος μας. Και θέλω να ρωτήσω ποιος θέλει να κάνει συγκεκριμένη όμως ερώτηση. Τζάκι Φώστερ, Πέτερ Φαντάλεν, Κλέρ Ντουίν, Γκεζίνε Μάισνερ. Παραμένουμε σε αυτό δύο λεπτά έκαστος για να ακούσουμε και την απάντηση. Την ομιλία σας θα μας τη δώσετε, ωραία, θα μας τη στείλετε και τις διαφάνειες για να μπορούμε να διαβάσουμε και τις λεπτομέρειες. Η Τζάκι Φώστερ. Δύο λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρένερ που ήρθε στην Επιτροπή μας ε, τόσο γρήγορα και είναι πάρα πολύ καθησυχαστικό αυτό ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία και με το Eurocontrol και με το ε, ΚΑΟ. Ε, περιέγραψε πάρα πολύ λεπτομερώς την κατάσταση για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή και πραγματικά χαίρομαι που λαμβάνετε σοβαρά υπόψη αυτό και ελπίζω να μην επαναληφθεί τέτοια τραγωδία, τέτοια καταστροφή, όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς εθέρες, ε, αλλά και ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ, Πέτερ Φαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, και σήμερα άκουσα τον κύριο Μπρένερ να μιλάει για την πρωτοβουλία ΙΚΑΟ και για το website για τα αλλαγή προφοριών στην ιστοσελίδα μεταξύ κρατών ε, εκτίμηση κινδύνου, ασφάλειας, θα το βελτιώσει. Με μεγάλους επένους το ανέφερε και ε, ότι περιμένει πολλά. Δεν είναι ο μόνος, το έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου μήνε επανειλημμένα. Εγώ διατηρώ πάρα πολλέ επιφυλάξεις για τους εξή δύο λόγους για αυτή την προσέγγιση. Πρώτον, ας υποθέσουμε 1η Ιουλίου του 2014, 17 ημέρες πριν ε, την κατάρριψη του αεροσκάφους ε, MH17. Ας υποθέσουμε ότι θα υπήρχε αυτή η βάση δεδομένων, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση ότι θα ήταν στο 300 ας πούμε και θα έκλεινε ε, ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας. Και η British Airways δεν πετούσε. Είχε άλλες προφορίες. Γιατί η KLM και η Lufthansa συνέχισαν τις πτήσεις τους πάνω από την Ουκρανία. Παρά το γεγονός ε, ότι δεν υπήρχε αυτή η βάση δεδομένων. Έστω, αν υπήρχε ε, την 1η Ιουλίου του 2014 θα μας βοηθούσε εγώ δεν με την αισιοδοξία σας. Και σε κάθε σελίδα, ό,τι βάζεις αυτό βγαίνει. Εξαρτάται από τα στοιχεία που εισάγει κανείς. Αυτή είναι η πρώτη μου επιφύλαξη. Δεύτερον, προηγουμένως είδα το χάρτη στην αρχή που μας έδειξε και η Κρυμαία ήταν ε, παρούσα στο χάρτη αυτό. Δεν την είχατε βγάλει. Τι γίνεται με την Κρυμαία, πετάτε από πάνω ακόμα, είναι λάθος το χάρτη αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιες είναι επικίνδυνες περιοχές εκτός της Ευρώπης κατά το Eurocontrol. Ξέρω ότι συχνά μιλάμε για την Συρία και τέτοια, αλλά και στην Αφρική υπάρχουν συγκρούσεις, στη Λιβύη. Δεκάδες ε, χιλιάδες κεφαλές και πύραυλοι ε, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς που είχε ο Καντάφη έχουν εξαφανιστεί. Ε, τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τους οπλισμούς και με αυτές τις περιφέρειες. Ευχαριστώ κυρία Κλούν. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρένερ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε για τους τελευταίους μήνες. Κάτι που μου έκανε εντύπωση όταν μιλήσατε για τις εκτιμήσεις κινδύνου και ασφαλείας για τα κράτη που συνεργάζονται τα λοιπά. Υπάρχουν κριτήρια, οι προδιαγραφές, οι πρότυπα και ποιος θα ορίζει αυτά. Για να υπάρχει ένα συντονισμός, κάποια κοινά κριτήρια. Μιλήσατε για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Αναφερθήκατε στο Τελαβίβ και πόσο χρήσιμα θα ήταν να υπήρχαν τέτοια δεδομένα. Πιο γρήγορα. Και για τους ε, Ρώσους και τα σχέδια πτήσης που υποβάλλουν, ε, πώς έχει γίνει αυτό, είναι πρόοδος λέτε, έχουν υποβάλει πρόσφατα τέτοια σχέδια, έχει προχωρήσει απλώς θεωρητικά. Ευχαριστώ, Γκεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Μπρένερ και από πλευρά μου πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, σύντομες. Πρώτον, είπατε ότι μπορεί να αποφασίσει μια αεροπορική εταιρεία αν θα πετάξει σε ένα διάδρομο ή όχι. Ε, ε, το αποφασίζει ο πιλότος. Ο πιλότος μόνο ή η οχι θα αποφασιζει ο πιλοτος ο πιλοτος μονο η η εταιρεια Ποιος είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο. Και δεύτερη ερώτηση για την εκτίμηση κινδύνου. Ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, υπάρχουν προδιαγραφές, ποιος το ορίζει αυτό. Και βλέποντας και προς το μέλλον, τι γίνεται με το Single European Sky, θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Ε, και έχω και εγώ ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Όλα αυτά ωραία και καλά εφόσον γίνουν. Αλλά ακούσαμε ότι η γερμανική κυβέρνηση ήδη ήξερε εκ των προτέρων ότι ήταν ε, ανασφαλές και επίφοβο να πετάει κανείς πάνω από την Ουκρανία. Και αυτό δεν το διαβίβασε ούτε στη Λουφτάνσα ούτε σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Τι κάνει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Μπορούμε να το ανεχτούμε, δεν ήταν ευθύνη της κυβέρνησης, δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης ή μπορεί μια κυβέρνηση ανεξαρτήτως πολιτικής ε, χρειάς να το κρατήσει για τον εαυτό της και να μην το μοιραστεί με κανέναν. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε, κύριε Μπρένερ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούει αγγλικά. I start with... Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, θα βοηθήσει βάσει βάση δεδομένων ρωτήσατε και αν θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τραγωδία τύπου της κατάρρευσης της πτήσης ε, MH17. Τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να μοιράζονται τα στοιχεία τους και την εκτίμηση κινδύνου. Αυτό είναι ήδη θετικό, γιατί μέχρι στιγμής δεν τους είχε ζητήσει κανείς να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να ρωτήσετε μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο τουλάχιστον στην Ευρώπη ή και πέρα από αυτή να υπάρχουν όχι μόνο συστάσεις αλλά κάπως ε, μια υποχρέωση, κάποια είδους υποχρέωση ε, ε, να μοιράζονται τις προφορίες. Στον ΙΚΑΟ αυτό είναι δύσκολο να γίνει, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλουμε να στραφούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς στο Eurocontrol έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα αρχίσαμε να συζητούμε το θέμα σε εθελοντική βάση για να δούμε αν υπάρχει αυτή η βούληση να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες ή αν είναι κάτι το ανεδαφικό που εμείς ζητούμε αλλά δεν το ακολουθεί κανείς ή παρά μόνο λίγοι. Προς το παρόν θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα κράτη. Ε, είναι πολύ χρήσιμη αυτή η σύσταση ΚΑΟ και μετά ε, να επανέλθουμε σε τέσσερις ή έξι μήνες για να δούμε ποια θα είναι η σύσταση και μπορεί τελικά να τελειοποιηθεί για να έχει και τα στοιχεία. Η κατάσταση νομίζω είναι διαφορετική. Είδαμε και την πρώτη συζήτηση μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Ε, υπάρχει ένα κράτος που δηλώνει ότι ένα αέριος χώρος του είναι ασφαλής και μετά βγαίνει ένα άλλο και λέει «Α, μην πετάτε οι δικές μου εταιρείε πάνω από την τάδε χώρα γιατί δεν είναι ασφαλής». Ε, βέβαια, μετά βγαίνει το πρώτο κράτος και διαμαρτύρεται. Και λέει από πού του βγάζετε αυτό το συμπέρασμα. Έχετε τέτοια σύσταση για το δικό μου ένα αέριο χώρο. Εγώ είμαι κυρίαρχο κράτος. Αλλά βάσει των διαφορετικών πληροφοριών που έχουν έρχονται δύο χώρες, τα συγκρίνουν και καταλήγουν σε ένα κοινό κείμενο το οποίο δεν έλεγε ότι είναι ασφαλές πλήρως να πετάει κανείς εκεί. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή τακτικής και συμπεριφοράς και όλο και περισσότερο Και αν δεν πετύχει θα έχω την ευκαιρία να έρθω να σας αναφέρω τι ίσως χρειάζεται περισσότερα. Προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Τα πρότυπα υπάρχουν στον ΙΚΑΟ, οι προδιαγραφές για το risk assessment που γίνεται η αξιολόγηση του κινδύνου. Και αυτό είναι υποχρεωτικό. Αν το κάνεις και είναι υποχρεωμένα τα κράτη να το πράττουν, θα πρέπει να ακολουθούν αυτή τη διαδικασία δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι είναι συγκρίσιμα αυτά. Το πρόβλημα ποιο ήταν στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα ε, της εκτίμησης αξιολόγησης κινδύνου δεν το, δεν το μοιράζονταν τα κράτη μεταξύ τους, δεν το διαβίβαζαν το ένα στον άλλο. Το πώς θα γίνει όμως αυτό και πώς διεξάγεται. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές προδιαγραφέ και πρότυπα από τον ΕΚΑΟ και είναι καθένα υποχρεωμένος να τα ακολουθεί. Για τα σχέδια πτήση, βεβαίως έχει δεσμευτεί η Ρωσία και σε υψηλό επίπεδο να τα ανακοινώνει. Το τελευταίο διάστημα είδαμε σωστά σχέδια πτήσης να υποβάλλονται και να διακινούνται. Μαθαίνει σιγά σιγά και η Ρωσία και η ρωσική αεροπορία να το κάνει πολεμική ε, το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουν ε, ε, τη βούληση. Όχι, ήταν θετική η προσέγγιση τους. Και τώρα είναι σε τεχνικό επίπεδο αυτό πώς τελικά οι διάφοροι οργανισμοί το βλέπουν αυτό. Αν δείτε τη διαφάνεια μου, είναι πολλές χώρες που έχουν κλειστό ένα αέριο χώρο γύρω από μας που είναι πολύ δύσκολο να μετακινούνται επιβάτες. Ε, από τη Συρία δεν ε, πετάει τίποτα και από τη Λιβύη. <laughs> Είναι λίγες οι χώρες σε σχέση με μια δεκαετία πριν γύρω μας ε, που έχουν τη δυνατότητα για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις αέριες ροές. Έχει περιοριστεί αυτός ο χώρος σε σχέση με λίγα χρόνια πριν και βεβαίως έχει αυξηθεί η εναέρια κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε ότι Βουλγαρία, Ρουμανία προς Τουρκία είναι μικρός ο διεύλος με πάρα πολύ μεγάλο φόρτο ε, και ροή. Αν υπήρχε κάποια τεχνική, ε, τεχνικό πρόβλημα που να εμποδίζει την ε, διέλευση θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Το ποιος αποφασίζει. Αν αποφασίσει ένα κράτος ότι τα αεροσκάφη που έχουν καταχωρηθεί στη χώρα ε, απαγορεύεται να πετάξουν πάνω από μια εναέρια, ε, σε ένα αέριο χώρο ε, μπορεί να το αποφασίσει η εταιρεία ή ο πιλότος. Μερικές φορές η εταιρεία το ρισκάρει, αλλά αν δεν το ρισκάρει ο πιλότος, ο πιλότος έχει τον τελευταίο λόγο Υπάρχει μια ιεραρχία στη λήψη των αποφάσεων, ε, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει όταν σου λέει χώρα μην πετά, σου λέει εταιρεία μην πετά. δεν μπορεί ο πιλότος να πει θα πετάξω. Ε, στον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό αν μας βοηθάει αυτό, μας βοηθάει για να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό, για να μοιραζόμαστε πληροφορίε σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας. Ε, ο ενιαίος ε, ευρωπαϊκός ουρανός ε, ήταν η κοιτίδα του διαχειριστή του χώρου, εσείς σε δική σας έμπνευση ήταν αυτή και είναι ένα καλό μέσο και εργαλείο που μπορούμε να το μεταξελίξουμε σε επίπεδο επιχειρησιακό για το μέλλον. Είναι ένα σημαντικό μέσων πριν από 30 χρόνια δεν υπήρχε, αλλά τώρα με τον όγκο που έχουμε στις αέρες μεταφορές και στην ε, κατάσταση ασφαλείας που έχουμε, δεν ε, μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε τη μετεξέλιξη αυτού του εργαλείου, γιατί είναι και μεγαλύτερες οι ανάγκες και οι απαιτήσει. Ελπίζω να απάντησα σε όλα. Δεν απαντήσατε στη δική μου ερώτηση όμως. Because Germany was informed. Δεν σας είπα ότι ήξερε η γερμανική κυβέρνηση για την Ουκρανία. Δεν μου απαντήσατε. Uh, uh, Α, μάλιστα ήταν δεν κατάλαβα τη γλώσσα λέει ο κύριος Βρένε, που με ρωτήσατε. Τι να σας πω. Είπα ε, στην ομιλία μου ότι ε, αυτό θα πρέπει να είναι το να ενημερώνει μια χώρα μόνο τις δικές της εταιρείες είναι μία Ευρώπη και μία ηρωή των πληροφοριών. Εγώ δεν ξέρω αν η Γερμανία είχε άλλη πληροφόρηση που δεν την ξέραμε εμείς κανένας άλλος. Όλα αυτά θα ήταν εικασίες. Αλλά με βάση τη νέα τώρα αντίληψη ενθαρρύνουμε τις χώρες να μοιράζονται τις πληροφορίες ε, σε αυτή την ιστοσελίδα μας, στον ιστότοπο χωρίς να αναφέρει την πηγή. Δεν λέμε ποιος το είπε, ε, αλλά ότι έχει την πληροφορία να τη μοιράζεται με τις άλλες χώρες και με τους ενδιαφερομένους για να μπορεί να χρησιμοποιείται αναλόγως και από άλλες εταιρείε. Υπήρξε ένα καλό παράδειγμα όπου λίγες χώρες στην Ευρώπη προχώρησαν και είπαν ότι θεωρούμε ότι είναι επισφαλές να πετά κανείς τις εξής ε, περιφέρειες. Και δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε την πηγή μας, αλλά έχουμε βάσιμες προφορίες, ωραία. Ε, να μας το πούνε. Και είχαμε και αντιδράσεις από την ελόγω χώρα που μας βοήθησε να βελτιώσουμε γενικότερα την κατάσταση ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την απάντηση όλων των ερωτήσεων και για την παρουσίαση και σας ευχαριστούμε. Και πάμε στο επόμενο θέμα και κλεισμένο των θυρών.